Ε, ε, welcome to Commissioner Θα καλωσορίσουμε την Επίτροπο Μπιενκόφσκα, αλλά προηγουμένως έχουμε δύο σύντομα σημεία. Η κυρία Μπιενκόφσκα θα περιμένει εκτός αίθουσας και ίσως να καπνίσει και ένα τσιγάρο, δεν ξέρω. Ε, φαντάζομαι πράγματα. Δεν μπορεί να μην ισχύει καν, θα τη ρωτήσω αργότερα. Λοιπόν, Επιτροπή, αποστολή της Επιτροπής Ήτρε στον Οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS την Πράγα 3 και 4 Νοεμβρίου 2015. Ενημέρωση. Τα τρία μέλη της Επιτροπής ε, Ήτρε επισκέφθηκαν τον οργανισμό του Ευρωπαϊκού GNSS, του Συστήματος Δορυφορικής Πλοήγησης, που ασχολείται και με, την, ε, με τα προγράμματα Γαλιλαίο και Έγνος και μας απασχολεί και η ασφάλεια των δικτύων εδώ και η ανάπτυξη της σχετικής αγοράς. Δείξαμε τη στήριξή μας προς το Γαλιλαίο ε, και τη σημασία που το αναγνωρίζουμε επιθυμώντας να είναι μία επιτυχία. Θα ήθελα λοιπόν τα μέλη της Επιτροπής Τη αποστολή αυτή να μας ε, ενημερώσουν. Ο συναδελφό Ρούμπικ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ ξεκινήστε την παρουσίαση. Έχετε το λόγο. Ε, sorry, President. Can you uh, again... με, με συγχωρείτε. Ποιο είναι το θέμα? Η αποστολή μας στο GNSS. να τονίσω ότι φυσικά αυτή ήταν η αποστολή που για πρώτη φορά έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτόν τον οργανισμό και αυτό το παγκόσμιο σύστημα πλοήγησης ε, θα είναι αποφασιστικό για την εξέλιξη των ευρωπαϊκών υποδομών. Το πρόγραμμα Κοπέρνικος ε, σχετίζεται άμεσα με αυτό και οι δορυφόροι, οπωσδήποτε, στο μέλλον θα προσφέρουν νέες δυνατότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία. Κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον και αποφασιστικό για μένα είναι η ακριβής μέτρηση του χρόνου που μπορεί να γίνει με αυτούς τους δορυφόρους σε πολύ λεπτομέρεια, σε μικρό επίπεδο. Αυτό το αξιοποιούμε για να υπάρχει ένα ευφυές δίκτυο, να υπάρχει απόλυτο συγχρονισμός των δικτύων στον τομέα του ηλεκτρισμού και επίσης ε, το αξιοποιούμε και για το νέο σύστημα 5G. Θα έχουμε λοιπόν καλύτερες επικοινωνίες, καλύτερα δίκτυα και κατά συνέπεια ευρύτερα η ψηφιακή ενιαία αγορά θα βασιστεί πολύ σε αυτά. Φυσικά αυτό το σύστημα το παγκόσμιο σύστημα δόρυφόρων παίζει πολύ ουσιώδη ρόλο και για την πλοήγηση. Υπάρχουν αλγόριθμοι που μπορούν να αξιοποιηθούν διαπιστώνουμε ότι περνάμε στην ιονή πραγματικότητα με αυτές τις δυνατότητες στην εικονική πραγματικότητα και αυτό μας ε, βοηθάει για να ιδρυθούν νέες εταιρείες στον τομέα αυτό. Υπάρχουν ε, ειδικοί όμιλοι επιχειρήσεων που δεν ε, παρέχουν μόνο τις βασικές υπηρεσίες, αλλά και περαιτέρω υπηρεσίες που αξιοποιούν τις υπηρεσίες αυτών των δορυφόρων σε συνδυασμό με σταθμούς επί του εδάφους που μας επιτρέπουν πολύ ακριβέστερες ε, μετρήσεις. Για παράδειγμα μπορούμε να μετρήσουμε καλύτερα πώς αναπτύσσονται τα δάση μας με διάφορους αισθητήρε τους οποίους μπορούμε να συνδυάσουμε και άρα προκύπτουν και νέες δυνατότητες για επιχειρήσεις, για επιχειρηματική δραστηριότητα. Και ήμουν και παρόν και στην διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προπολογισμό και διαπιστώσαμε ότι γίνονται περικοπές σε αυτούς τους δύο τομείς. Η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι δεν είναι αναγκαίες όλες οι πληρωμές που προβλέπονταν για το 2016, αλλά οι υποχρεώσεις παραμένουν όσες ήσαν, ούτως ώστε το 2018 θα είναι διαθέσιμες οι πιστώσεις που θα πρέπει να εκταμιευθούν. Οπότε, ίσως να υπάρξει και συμπληρωματικός προπολισμός για το 2016 για τα συστήματα αυτά. Η Επιτροπή έχει εμπιστοσύνη ότι θα μπορέσει να στηριχθεί δημοσιονομικά, δημοσιονομικά αυτή η προσπάθεια και ο οργανισμός αυτός μας είπε ότι έχει έλλειψη προσωπικού ήδη. Ξέρετε ότι έχουμε στόχους να μειωθεί το προσωπικό μας ε, στην ε, Ένωση. Όμως εμείς τονίσαμε ότι για τον οργανισμό αυτό πρέπει να αυξηθεί το προσωπικό. Είναι αναγκαίο αυτό. Και πιστεύω ότι όταν θα δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια του χρόνου, όταν θα αποδειχθεί πόσο χρήσιμα είναι όλα αυτά και ότι μέχρι το 2020 θα έχουν πλήρως αναπτυχθεί, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε ένα συνδυασμό του τομέα αυτού με τις άλλες οργανώσεις και οργανισμούς του τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Να παρακαλέσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους που πήγαν στην Πράγα, τον κύριο Τζανονάτο και τον κύριο και αν θέλουν να προσθέσουν κάτι. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να προσθέσω σε αυτά που είπε ο το εξή. Σήμερα στον πλανήτη λειτουργούν δύο συστήματα γεωγραφικού ε, γεωγραφικής πλοήγησης. Το ένα είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και στην Ευρώπη, το GPS, και το άλλο είναι αυτό της Ρωσίας. Δημιουργήθηκαν για σκοπούς άμυνας, αλλά μετά εξελίχθηκαν σε εφαρμογές προς όφελος των πολιτών, μη δηλαδή δηλαδή χρήσεις, ε, των οποίων αποφελούμαστε κι εμείς. Τα συστήματα αυτά γεωγραφικής πλοήγησης ε, έχουν εξέλιξη και στην Κίνα και στην Ινδία. Επίσης υπάρχει και το δικό μας σύστημα, το Galileo, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2019. Το σύστημα Galileo θα έχει το επιπλέον χαρακτηριστικό ότι θα μπορεί και να λαμβάνει δεδομένα από όσους βρίσκονται ε, στην ε, επιφάνεια της γης, οπότε θα μπορέσει να συμπληρώσει τα υπάρχοντα συστήματα. Κάτι που δεν επιτρέπουν τα συστήματα αυτά, το GPS και το ρωσικό συστήμα. Ε, υπάρχουν τουλάχιστον 30 δορυφόροι βέβαια που θα χρειαστούν, 6 ως το τέλος της χρονιάς. Το σύστημα, όπως είπα, θα ολοκληρωθεί το 2019. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη και έδειξε πώς έχουν προχωρήσει οι προσπάθειες ε, δημιουργίας αυτού του συστήματος που θα δώσει και στην Ευρώπη τη δυνατότητα να συμμετάσχει πλήρως στο παγκόσμιο αυτό εγχείρημα. Πέραν αυτών είδαμε και τι γίνεται με το Κοπέρνικο, σύστημα φωτογράφησης του πλανήτη που επιτρέπει με απόλυτη ευκρίνεια να δούμε και την κατάσταση του περιβάλλοντος ε, σε, πολλά σημεία, σε όλα τα σημεία του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, φωτογραφίσεις υψηλής ευκρίνειας και υπάρχει και το σύστημα έγνος που είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τα μικρά αεροδρόμια εκεί που τα αεροσκάφη για να προσγειωθούν όταν δεν υπάρχει καλή ορατότητα ή μηδενική ορατότητα χρειάζονται πολύ συγκεκριμένη γεωγραφική καθοδήγηση για να ξέρουν ακριβώς πού βρίσκονται. Συνολικά η επίσκεψη ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ πλούσια και μας δέχτηκαν με πολύ μεγάλη εγκαρδιότητα. Να επιφεληθώ για να πω και κάτι ακόμη. Οι υπάλληλοι, όσοι εργάζονται για τον Καλλιλέο, το σύστημα αυτό αναζήτησης που ε, μελετάτε στην Πράγα λαμβάνουν τέτοιους μισθούς που δυστυχώς δεν έχουν καλό κίνητρο για να παραμείνουν εκεί. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς πρέπει να διορθωθεί ο μηχανισμός μέσω του οποίου προβλέπουμε τις αμοιβέ αυτών των ερευνητών, διότι μετά από κάποιο μικρό διάστημα ψάχνουν διαφορετική λύση για την καριέρα τους. Ο επικεφαλής του προγραμματός είναι διαθέσιμος για να έρθει εδώ και να μας μιλήσει όχι μόνο για τους μισθούς, αλλά να μας παρουσιάσει και το εγχείρημα αυτό γενικότερα. Θα ήταν καλή ιδέα λοιπόν να τον φιλοξενήσουμε, να τον δεχθούμε κάποια στιγμή εφόσον το αποφασίσουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε για αυτή την πρόταση. Συνάδελφε το Σανόσκι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα συμπληρώσω απλώ όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ήταν ε, πραγματικά εντατική η επίσκεψη γιατί ένα μισάωρο, ένα τέταρτο, είχαμε νέου ομιλητέ, νέου εισηγητέ και πραγματικά δεχτήκαμε σωρία πληροφοριών. Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά και για την Επιτροπή μας μεταξύ άλλων. Ο οργανισμός αυτός συνάπτει συμβάσεις ε, σημαντικότατης αξίας, δισεκατομμυρίων ευρώ και η όλη επιχειρηματική δραστηριότητα που αφορά τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης θα γνωρίσει διπλασιασμό της εμπορικής της αξίας τα επόμενα χρόνια. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα συστήματα αυτά που μας παρουσιάστηκαν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Επιτρέπουν να ε, έχουμε και μεγαλύτερη ασφάλεια σε πολλές περιπτώσεις, κάτι που αυτή τη στιγμή είναι και θέμα επικαιρότητα. Ε, το πρόγραμμα Κοπέρνικος για την ώρα δεν είναι τόσο καλά προστατευμένο και δεν ενισχύεται τόσο καλά όσο το Γαλιλαίο, αλλά θα συμφωνήσω με αυτά που είπε και ο συνάδελφος Ντανονάτο. Ε, είναι σημαντικότατα όλα αυτά, πρέπει να τους δώσουμε την ανάλογη προσοχή Και να μην ξεχνάμε ότι στην Πράγα οι μισθοί δυστυχώ είναι αποθαρρυντικοί. Οι ερευνητέ δεν έχουν επαρκέ κίνητρο για να παραμείνουν εκεί. Κάτι λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη θέση μα. Θα κλείσω εδώ την παρέμβασή μου. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για τι τοποθετήσει σα. Ευχαριστώ και για την επίσκεψη και για την ενημέρωση. Νομίζω όλες οι παρατηρήσεις θα πρέπει, νομίζω ότι όλες αυτές μάλλον οι παρατηρήσεις θα πρέπει να μας απασχολήσουν στις συζητήσεις μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη όσο μας είπατε και θα φροντίσουμε να αποστείλουμε τα ανάλογα μηνύματα τη φυλακή και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών. Μιλήσαμε για, την, για τον οργανισμό δορυφορικής πλοήγησης στην Πράγα. Πάμε τώρα στο σημείο 9. Αποστολή της ΙΤΡΕ στο 10ο συνέδριο του Φόρουμ Διαδικτυακής Διακυβέρνησης. Μία ε, επίσκεψη στη Βραζιλία με αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων. Από τέσσερα μέλη που είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν πέρσι φτάσαμε τους 9 φέτος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε επίσκεψη κάθε χρονιά στην ετήσια αυτή ε, συνέλευση του Φόρουμ Διαδικτυακής Διακυβέρνησης. Η Επιτροπή μας, ΙΤΡΕ είναι η καθήλυνα αρμόδια για τα θέματα αυτά. Ναι, είναι η Επιτροπή που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Οπότε είναι σημαντικό να αναλαμβάνουμε και την ευθύνη για την παρακολούθηση των θεμάτων αυτών. Εννέα λοιπόν μέλη από πολλές διαφορετικές επιτροπές συμμετείχαν, αλλά κυρίως ε, η δική μας επιτροπή ήταν αυτή που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο επικεφαλής της αποστολής στο συνέδριο της, ε, του Φόρουμ Διαδικτυακής Διακυβέρνησης στο Ζουάου Πεσόα στη Βραζιλία ήταν ο συνάδελφος Ζουρίνιου. Σας δίνω τρία λεπτά για να μας πείτε τι έγινε στη Βραζιλία πριν από λίγες εβδομάδες. Σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι δύσκολο να τα ανακεφαλαιώσω όλα σε τρία λεπτά. Όπως είπατε, η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, της οποίας είχα την τιμή να προεδρεύω, εξονόματος της Επιτροπής μας, ήταν η μεγαλύτερη και η πιο αντιπροσωπευτική από ποτέ. Τέσσερις επιτροπής, Ήτρε, Κούλτ, Λίμπε και Γιούρι, με την συμμετοχή της ΣΤΟΑ, δηλαδή τεχνολογική υποστήριξη και μεγάλη στήριξη από τις πολιτικές ομάδες. Είχαμε πάντοτε υπόψη την εντολή που μας ανατέθηκε. Εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ένα ψήφισμα για την συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο μέλλον αυτού του φόρου. Την ε, παρουσία μας τη με την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με προκαταρκτικές ε, συνεδριάσεις, με την παρουσία του Επιτρόπου Άνση που ήταν εκείνος που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φροντίσαμε να υπάρξει παράταση της εντολής του διαδικτυακού φόρουμ, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να έχουν αποτελεσματική δράση για τη χρηματοδότηση και το μοντέλο που χρησιμοποιείται και είχαμε μια πολύ σημαντική συζήτηση στο φόρουμ. Δηλαδή να δούμε κατά πόσον η πολυμερής προσέγγιση είναι προτιμότερη από τις πολυετερικές σχέσεις. Προσπαθήσαμε επίσης να συνεισφέρουμε στην σαφή τοποθέτηση στήριξης των δράσεων για το διαδίκτυο για τις δράσεις και τα ονόματα, να υπάρχει ένα ελεύθερο διαδίκτυο, εύκολα προσβάσιμα. Είχαμε πολλές διμερείς συνομιλίες όπως αναφέρεται στο έγγραφο που ήδη έχουν λάβει οι συνάδελφοι, και τα θέματα που πλέον συζητήθηκαν πέραν του μοντέλου διακυβέρνηση για το διαδίκτυο ήταν αυτά που τα συζητούμε καθημερινά εδώ στο Κοινοβούλιο όταν συζητούμε την ψηφιακή ατζέντα. Μερικά θέματα μάλιστα ήταν ακόμη πιο δημοφιλή στο φόρουμ λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. Η οικονομία του διαδικτύου, η πρόσβαση και η πολιτιστική επικοινομορφία στο διαδίκτυο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η ελευθερία στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, πώς να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές με ασφάλεια και προστασία, πώς να υπάρξουν νέες πρακτικές στο θέμα λόγου χάρη του zero rating για να προσελκύσουμε και νέους χρήστες. Η κοινή θέση Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντικατοτρίζεται στο τελικό έγγραφο που προέκυψε από το Φόρουμ Διαδικτυακής Διακυβέρνησης και συμπεραίνω ότι γενικώ η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Ευρωκοινοβουλίου ήταν πάρα πολύ σκόπιμη. Θα πρέπει να ε, παραμείνουμε, να, να συνεχίσουμε να δίνουμε προσοχή στην συμμετοχή όλων στα θέματα που αφορούν το διαδίκτυο ως προς τη διακυβέρνησή του και Επιμένω εδώ ότι θα πρέπει πρωταγωνιστικό ρόλο στο συντονισμό να έχει η Επιτροπή μα, ήτρε. Διότι τα θέματα αυτά είναι απλά και εκεί που μπορεί να δώσει κάποιο προστιθέμενη αξία είναι ακριβώ η Επιτροπή μα. Και κλείνοντα, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω όλου του συνεργάτε που μα συνόδευσαν. Ήταν πολύ αποτελεσματική η στήριξή του και του συναδέλφου από άλλε επιτροπέ, χάρη στου οποίου σχηματίσαμε μια αντιπροσωπεία που έφερε εις πέρας νομίζω άριστα την εντολή που, την, ε, που είχαμε την τιμή να αναλάβουμε από εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μας είπατε. Τέσσερις συνάδελφοι από τον... Ε, βλέπω ότι ε, ήταν από, τις, από την Επιτροπή μας και πέντε από τις υπόλοιπες. Ε, πολιτισμού, πολιτικών ελευθεριών κλπ. Οπότε όλοι μαζί ήμασταν συνυπεύθυνοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους εννέα συναδέλφους. Ε, δύο συνάδελφοι εδώ παρόντες. Είναι και η κυρία Καϊλή εδώ. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μήπως θέλετε να προσθέσετε κάτι κυρία Καϊλή. Έχετε το λόγο. thank you, Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα απλώ να μοιραστώ κάποια σκέψη μαζί σα και να ευχαριστήσω την γραμματεία, ειδικότερα τον Ήγκο, για την καταπληκτική του δουλειά, γιατί πραγματικά τα πάντα είχαν συμπεριληφθεί ε, για ολόκληρη την ημέρα. Ε, το, η Ζωάο είναι η τέταρτη πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο. Εμείς δεν αισθανόμασταν πάντως ότι ε, ήμασταν σε κίνδυνο, αισθανόμασταν πολύ ασφαλείς. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί νομίζω ότι είχαμε σημαντικότατες ε, συναντήσεις από τις μεγάλες εταιρείες που ε, συμμετείχαν. Να ευχαριστήσω και τον Κάρλος γιατί ηγήθηκε όλης αυτής της αντιπροσωπείας ε, δεν είχαμε καθόλου ελεύθερο χρόνο, ήταν ε, όλα οργανωμένα. Τα ζητήματα που συζητήσαμε, κυβερνοασφάλεια, ε, ε, το θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου. Όλα ήταν πολύ ενδιαφέροντα θέματα και ήταν πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον το ότι μπορέσαμε να εκφράσουμε την άποψή μας και στους υπόλοιπους εταίρους που συμμετείχαν σε αυτό το φόρουμ. Ο αντιπρόεδρος ήταν εκεί, αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, της Βραζιλίας και νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι όλος ο κόσμος φοβάται το κοινοβούλιο και την επιπλέον ρύθμιση, αυτό είναι πολύ ε, σημαντικό. Υπάρχει και στην ενημέρωση το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης. Ε, συζητήσαμε με διάφορες χώρες, όπως για παράδειγμα στην Ινδία, ε, κατεβάζουν sites που βοηθούν τα παιδιά και προσπαθούν να προωθήσουν τη σωστή χρήση του ίντερνετ Νομίζω λοιπόν ότι οι χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό και θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να είναι δημοκρατικός ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Και όπως είπε και ο Κάρλος, ελπίζουμε να συνεχιστεί η προσπάθεια αυτή. Ε, ελπίζουμε να μπορέσουμε να συμμετέχουμε και του χρόνου δεδομένη τη εξαιρετική εργασία τη γραμματεία μα, είμαι βέβαιη ότι η συνέχιση τη διαδικασία αυτή ε, θα γίνει πάρα πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχαριστώ και για την παρουσία σα στη Βραζιλία. Περνάμε τώρα στο σημείο 10 τη ημερήσια διάταξη. Ε, θα ήθελα να ε, ζητήσω συγγνώμη από την Ελισπιέτα Μπιενκόφσκα, την Επίτροπο. Έχουμε καθυστερήσει 5 λεπτά. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Μπενκόφσκα. η Επίτροπος ε, ε, Εσωτερικής Αγοράς Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας. Ε, θυμάμαι τα πάντα, αλλά θυμάστε εσείς πολύ περισσότερα. Η ανταλλαγή απόψεων είναι τμήμα του διαρθρωτικού διαλόγου μας και είναι μια ευκαιρία για όλους τους ευρωβουλευτές να θέσουν ερωτήματα για ένα πολύ σημαντικό θέμα το πρόγραμμα εργασίας τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το επόμενο έτος θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα προτείνεται. Κυρία Επίτροπε, για την επόμενη χρονιά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι καλύτερη νομοθεσία σημαίνει και ευθύνη για μας είναι ε, ιδιαίτερα σημαντική αυτή η διάσταση για όλους τους τομείς και όλος ιδιαίτερος για την ε, εσωτερική αγορά. Είμαστε εμεί όλος ιδιαίτερος μάλιστα υπεύθυνοι για την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι δική μας ευθύνη. Με μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν περιμένουμε την ε, ανταλλαγή απόψεων με σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι ε, ευρωβουλευτές, ε, όπως σωστά υπόθηκε είναι τμήμα του διαρθρωμένου διαλόγου η σημερινή μας συνάντηση. Σας έχω υποσχεθεί να σας τηρώ ε, ενήμερους, αλλά ένα σημαντικό τμήμα της σημερινής μας συνάντησης. Ελπίζω ότι θα είναι σημαντικότερο και πιο ενδιαφέρον από τη δική μου παρουσίαση. Θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα για τη στρατηγική, για την ενιαία αναφορά, μετά για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα ζητήματα Volkswagen και τα ζητήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως επίσης και για τα σχέδιά μας για το επόμενο έτος, στο πλαίσιο αυτό, γιατί όπως υπόθηκε, αυτά είναι δύο σημεία τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν με τη στρατηγική για την ενιαία αγορά. Έχουμε επικεντρωθεί σε, τρία βασικά ε, αποτελέσματα. νέε ευκαιρίες για τους καταναλωτές, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Εξυγχρονισμός της βιομηχανίας μας ε, και της οικονομίας μας γενικότερα. Και κατά την άποψή μου το σημαντικότερο τμήμα της στρατηγικής ε, όλα αυτά είναι σημαντικά βεβαίως, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το, το θέμα της αποτελεσματικότητας, η δημιουργία ευκαιριών, δηλαδή νέες ευκαιρίες ε, για τους καταναλωτές μας, για τους επαγγελματίες μας, για τις επιχειρήσεις μας, όπως επίσης και για τις νέες επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε θέσει τα θεμέλια με την πρότασή μας για την Έναση κεφαλαία αγορών. Είχαμε πει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα της ευρύτερης ε, εικόνας που θέλουμε ε, να, ε, να προτείνουμε ως στρατηγική. Είναι κάτι που πρόκειται να εγκριθεί αύριο. Είναι το θέμα της, του πακέτου της κυκλικής οικονομίας για το οποίο είμαι υπεύθυνη από κοινού με τον Πίτροπο Βέλα. Εμείς ε, θα παρουσιάσουμε ένα συντονισμένο σύνολο μέτρων ε, και δράσεων για να δούμε πώς μπορούμε να ε, μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Είναι κάτι που δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το τμήμα της στρατηγικής μας πρέπει κατά τη διάρκεια της περίοδου εφαρμογής να το επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο γιατί τότε θα το συνοδεύσουμε με πολύ λεπτομερές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δράσεις για την εφαρμογή εφαρμογή. Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις θα προτείνουμε, μέτρα για δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηματίες. Ε, ήταν ένα από τα ε, αιτήματα που ε, μας ε, επαναλάμβαναν ε, συνεχώς οι επιχειρήσεις, οπότε αποφασίσαμε να δώσουμε στους επιχειρηματίες ε, μία δεύτερη ευκαιρία. Κάτι ακόμη πάρα πολύ σημαντικό, σαφή καθοδήγηση για το πώς οι κανόνες και η φυστάμενη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει στη συνεργατική οικονομία, γιατί είμαι βέβαιη ότι πρέπει να έχουμε μία ενοποιημένη προσέγγιση προσέγγιση προς την κατεύθυνση της συνεργατική οικονομίας, όχι όπως έχουν τα πράγματα τώρα που είναι εντελώς διαφορετικά τα σύνολα των ε, ε, μέτρων και διαφορετικές προσεγγίσεις ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Ένα δεύτερο σύνολο αποτελεσμάτων να έχουμε ένα ενημερωμένο σύστημα προδιαγραφών, δηλαδή να έχουμε αποτελέσματα σύντομα, άμεσα και να δώσουμε μεγαλύτερη ε, πρόσβαση ε, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως. Και το τρίτο θέμα είναι η ε, ύπαρξη αποτελεσμάτων, όπως είπα, κυρίως καθοδήγηση και κανόνες, κανόνες και καθοδήγηση για το πώς θα εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Επιτόπου προτείνουμε λοιπόν μια ευφυή στρατηγική επιβολής, ε, ενημέρωση και αναβάθμιση της ε, εποπτείας της αγοράς ε, αγαθών και υπηρεσιών και θα ήθελα να σας πω και ορισμένα πράγματα για τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις εκπομπές ρήπων στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής πρέπει να τονίσω και πάλι και δεν μπορώ να το τονίσω αρκετά πόσο σημαντικό είναι να ε, υπάρξει αναβάθμιση ε, των ε, υπηρεσιών, της αγοράς υπηρεσιών μας. Πρέπει να αντιδράσουμε συλλογικά και άμεσα, γιατί όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε εξουσία εκτέλεσης των κανονισμών σε εθνικό επίπεδο, όμως εγώ ανέλαβα πρωτοβουλία ε, αυτή τη στιγμή διερευνούμε σε εθνικό επίπεδο, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και ελπίζω ε, κατά τις επόμενες ημέρες να έχουμε τα αποτελέσματα γιατί η προθεσμία ήταν εχθές, η προθεσμία που ε, μας είχε δώσει η Volkswagen για τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής και δεύτερον, δύο ακόμη σημαντικά ε, θέματα, η βελτίωση της δοκιμής σε πραγματικές συνθήκες για την εκπομπή ρήπων έγινε συζήτηση σε μια ρυθμιστική Επιτροπή και κατά τη δική μου άποψη υπήρξε ένας καλός συμβιβασμός. Ήταν απαραίτητο να υπάρξει ε, ένας συμβιβασμός γιατί χρειαζόμαστε ε, μία ε, αξιόπιστη διαδικασία δοκιμών γιατί θέλουμε να μειώσουμε από 400 ε, μιλιγκράμμα ανά χιλιόμετρο σε 160 ε, τις εκπομπές και ελπίζουμε ότι η νέα διαδικασία θα μας βοηθήσει μέσα σε δύο χρόνια να το καταφέρουμε αυτό. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να υπερψηφίσετε την πρόταση αυτή γιατί αυτός ο συμβιβασμός κατά την άποψή μου είναι ένας καλός συμβιβασμός, ο οποίος ε, αποτελεί μία ισορροπία μεταξύ της περιβαλλοντικής πτυχής και από την άλλη είναι εφικτός για τη βιομηχανία. Είναι φιλόδοξος στόχος, αλλά εφικτός. Τρίτον, ε, νέες ε, διαδικασίες δοκιμών για τη μέτρηση κατανάλωσης καυσίμων. Το επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ο Επίτροπος Κανιέτε είναι ο ε, Επίτροπος ο οποίος είναι υπεύθυνο για το ε, θέμα αυτό. Ελπίζουμε να έχουμε τα αποτελέσματα στους επόμενους μήνες. Κάτι ακόμη πολύ σημαντικό, πρόταση ενίσχυσης ε, της έγκρισης τύπου και της ανεξάρτητης διαδικασίας δοκιμών των οχημάτων. Οι προτάσεις μας οι λεπτομερείς θα είναι έτοιμες κατά τη διάρκεια του ε, Δεκεμβρίου. Όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, πρέπει να είμαστε πραγματικά ε, ταχύτατοι. Εδώ η στρατηγική της ενιαίας αγοράς θα μας βοηθήσει. Δεύτερο σημείο που αφορά την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Η προσέγγιση την οποία ε, έχουμε ακολουθήσει στη στρατηγική μας ε, είναι οι 22 δράσεις ε, για τρία αποτελέσματα, ανάπτυξη και απασχόληση, όπως επίσης και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μας. Ελπίζουμε ότι κατά τον επόμενο μήνα θα παρέχουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Χρειαζόμαστε βέβαια και τη δική σας άποψη. Γι' αυτό η σημερινή τόσο σημαντικές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτά να ε, συνάδουν με τις υπόλοιπες στρατηγικές μας, όπως για παράδειγμα τη στρατηγική για την ψηφιακή αγορά. Ε, είναι εξίσου σημαντικό και αυτό. Ε, η ψηφιακή αγορά, η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και τον εξυγχρονισμό της βιομηχανίας μας που είναι ένα πολύ ευρύτερο θέμα. Τον Ιούνιο αναφέρθηκα σε μία πρόταση για ε, την βιομηχανική ανταγωνιστικότητα. Είναι ένα βασικό θέμα η στρατηγική για την ενιαία αγορά προκειμένου να υπάρξουν αποτελέσματα στο πλαίσιο αυτό. Να σας δώσω τρία παραδείγματα ένα σύστημα εξυγχρονισμένο ε, τυποποίησης, κάτι το οποίο θα μας δώσει κρινόμαστε γρήγορα σε αλλαγές στην αγορά και θα το καταστήσει ευκολότερο στις εταιρείες να συμμετέχουν σε μια ε, ευρύτερη ε, αλυσίδα ε, παραγωγής και κατανάλωσης και νομίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο ε, θα μας δώσει τη δυνατότητα να ε, διευκολύνουμε ακόμη περισσότερο τα μέτρα αυτά είναι, ε, είναι πολύ ευρύτερο το θέμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ τώρα. Θέλουμε να αναφερθούμε σε βασικά προβλήματα τα οποία πλήττουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως για παράδειγμα την έλλειψη επενδύσεων, τις ενεργειακές τιμές, τους πόρους την αποδοτικότητα και τις αθέμητες πρακτικές. Όλα αυτά τα θέματα θα τα, ε, θα τα ε, επεξεργαστούμε κατά το επόμενο έτος να σας πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά την άμυνα και το διάστημα, γιατί είναι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες ε, που εντάσσονται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016. Για το διάστημα θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμα, ε, τη στρατηγική μας για το διάστημα με τις προτεραιότητες και τους στόχους μας. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των προγραμμάτων Κοπέρνικος και Γαλιλαίος για το διάστημα. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία επιταχύνουν συνεχώς και ε, τα οποία λειτουργούν, λειτουργήσαν καλά κατά τη διάρκεια του 2015. Ε, θέλουμε λοιπόν να τους δώσουμε όλες τις ευκαιρίες, να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό τους, θέλουμε να ενισχύσουμε ε, καλύτερη απορρόφηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των προγραμμάτων αυτών και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις αλλαγές την ε, παγκόσμια αλλαγή των προγραμμάτων για το διάστημα και να έχουμε μια ευρωπαϊκή απάντηση σε όλα αυτά. Παρά το γεγονό ότι είναι πολύ νωρί ακόμη να παρουσιάσω λεπτομέρειε, υπάρχουν κάποιε προτεραιότητε. Το συζητήσαμε χθε ε, στο πλαίσιο τη Προεδρία του Λουξεμβούργου. Ε, νομίζω ότι πρώτα πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρω τα προγράμματα Γαλιλαίος και Κοπέρνικος, να ε, μπορέσουμε να ενισχύσουμε την απορρόφηση στην αγορά από τις δημόσιες αρχές ε, των προγραμμάτων αυτών και των αποτελεσμάτων και επίσης να δούμε τι εργαλεία πολιτικής χρειαζόμαστε για να υπάρξουν νέες ευκαιρίες στην αγορά και να δούμε επίσης ε, και θέματα όπως η πρόσβαση ε, στο ε, διάστημα, να υπάρξουν περισσότερες προτεραιότητες, όπως επίσης να υπάρξει και καλύτερο πλαίσιο. Μπορεί να μην είναι το σημαντικότερο θέμα, αλλά πρέπει να υπάρχει σωστή διαχείριση. Όσον αφορά την άμυνα, που είναι επίσης ε, εν μέρη συνδεδεμένο με το θέμα της διαστημικής πολιτικής, ε, θα ε, εγκρίνουμε το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Άμυνας με δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, την ενίσχυση το, της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, όπως επίσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας το πρόγραμμά μας ε, έχει να κάνει με την άμυνα, με την έρευνα, ε, την ενίσχυση ε, των δυνατοτήτων και των τεχνολογιών. Επίσης προσπαθούμε να ενσωματώσουμε υπάρχουσες προτεραιότητες και το πρόγραμμα αυτό θα συνάδει με την ενίσχυση άλλων πολιτικών όπως για παράδειγμα την ενίσχυση της, πολιτικής, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας Επίσης, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, θα κατατεθεί μια νέα πρόταση για ε, τη δορυφορική ε, επικοινωνία ε, μεταξύ μεταξύ των κυβερνήσεων. Όλα αυτά, λοιπόν, θα ε, γίνουν την επόμενη χρονιά. Εγώ θα σας ενημερώνω και κατά τη διάρκεια της επόμενης ε, χρονιάς. Ο στόχος μας είναι να υπάρξουν οι συνθήκες για την ανάπτυξη, για την ύπαρξη θέσεων απασχόλησης, αλλά ε, επίσης και για την ενίσχυση της βιομηχανίας μας, της βιομηχανίας μας και της ανταγωνιστικότητάς της. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσίασή σας. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε, έλεγα, τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Ο Σνάλφος Χάριντς, από πλευράς του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Με συγχωρείτε που χρειάστηκε να βγω. Χτύπαγε πολύ δυνατά το τηλέφωνό μου. Με συγχωρείτε γιατί ήμουν λίγο αγενής. Να δούμε λίγο ευρύτερα το θέμα. Είστε υπεύθυνοι για τη βιομηχανία ως Επίτροπος. Έχω αυτό το σκάνδαλο. Ε, μιας πολύ σημαντικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Πολύ σημαντικής για την ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία για τις τεχνολογίες μας, για τις τεχνολογίες των κινητήρων diesel. Ακούμε επίσης ότι το πρόβλημα είναι οι κινητήρες diesel. Πρέπει να τους καταργήσουμε, να περάσουμε σε ηλεκτρικούς κινητήρες. Αλλά η Ευρώπη έχει εδώ ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Είναι στην ακμή της τεχνολογίας οι κινητήρες αυτοί. Άρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον μας. Καταλαβαίνω πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκές δομές, αλλά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς μπορείτε να παίξετε έναν ε, πολύ σημαντικό ρόλο και προβεβλημένο. Πώς σκοπεύετε να υπερασπιστείτε τη βιομηχανία μας, πώς θα στηρίξετε, πώς θα ενθαρρύνετε την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι μόνο θέμα Volkswagen. Αυτή είναι μια ευρύτερη απόπειρα που ε, ξεκινάει από τους ανταγωνιστές μας. Και πώς θα το συνδυάσετε με τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές μας για τις εκπομπές. Ευχαριστώ από πλευράς ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο συνάδελφος Νίκα. Ευχαριστώ. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τη Ρουμανία, λέει και ο Πρόεδρος. Είναι η εθνική Ορτή της Ρουμανίας. Όπως είπα και προηγουμένως, ε, συγγνώμη Ντάν, δεν επανέλαβα αυτό που είπα στους συντονιστές, ότι είναι σήμερα η εθνική Ορτή της Ρουμανίας. Σήμερα είμαστε όλοι Ρουμάνοι, μπορείτε να μιλήσετε ε, ρουμανικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Η Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο προσπαθούν να ε, προωθήσουν τα συμφέροντα της βιομηχανίας. Και είναι σημαντικό μαζί μας να συζητήσετε πώς θα επιτύχουμε ανάπτυξη γιατί υπάρχει κάποια σύγχυση. Δεν λαμβάνουμε πάντα την αναγκαία πληροφόρηση που χρειαζόμαστε και δεν λαμβάνουμε πάντα την πληροφόρηση από τους αρμόδιους, για παράδειγμα την Γενική Διεύθυνση Growth. Δεν καταφέραμε να αποφασίσουμε μια έκθεση γιατί δεν είχαμε την αναγκαία πληροφόρηση, για παράδειγμα. Η Γενική Διεύθυνση Growth ε, βεβαίως εκπροσωπείται από το Γενικό της Διευθυντή αλλά ήρθε και μα είπε αυτός ο Γενικός Διευθύντης ότι η αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η Γενική Διεύθυνση ε, ΚΛΙΜ. Κανείς δεν ήθελε βεβαίως να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο γενικών διευθύνσεων. Δεν έχουμε για παράδειγμα ακόμη την έκθεση για τις επιπτώσεις του ETS στην βιομηχανία. Πολύ λίγη πληροφόρηση έχουμε και για τις ερωτήσεις που θέσαμε δεν λάβαμε καμία απάντηση. Μας είπαν ότι ίσως σήμερα το απόγευμα. Χθες κάναμε μια συζήτηση για τον τομέα της ενέργειας. Η Γενική Διεύθυνση Ενέργεια βέβαια θα έπρεπε να είναι αρμόδια. Και ένας εκπρόσωπος της, αν κατάλαβα καλά, μας είπε ότι ο κλάδος ε, βεβαίως ε, απασχολεί ιδιαίτερα αλλά είναι κυρίως θέμα αρμοδιότητας Γενικής Διεύθυνσης Growth. Τίθεται λοιπόν θέμα πραγματικά αξιοπιστίες, γιατί ο κλάδος πρέπει να ξέρει ποιο το πλαίσιο για να μπορεί να κάνει μακροπρόθεσμη ε, προσπάθεια σχεδιασμού. Δεν είναι δυνατόν οι τιμές να αλλάζουν από την ε, μία μέρα στην άλλη. Για παράδειγμα, έχουμε τα εφή δίκτυα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει να αλλάζουν οι τιμές, να μεταβάλλονται, να μειώνονται, να αυξάνονται. Είναι πολύ δύσκολο για την ε, βιομηχανία μας. Αυτή είναι η προσέγγιση υπό την οποία εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιομηχανία μας. Νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε, γιατί μπορεί τελικά να καταστρέψουμε τη βιομηχανία μας. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πώς καθορίζουμε τη στρατηγική μας. Θεωρώ λοιπόν ότι οι αρμόδιοι της Γενικής Διεύθυνσης Growth θα έπρεπε να είναι παρόντες. Δεν είναι δυνατόν οι τιμές να αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχετε συνεκτική στρατηγική και σας ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Ευχαριστώ. Για το ECR, μήπως είναι και η εθνική γιορτή της ε, Τσεχικής Δημοκρατίας, όχι παρόλα αυτά μπορείτε να μιλήσετε τσεχικά. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πρέπει να επιβεβαιώσω ότι δεν είναι σήμερα η εθνική μας εορτή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να μιλήσω ρουμανικά. Οπότε θα μιλήσω τσεχικά. Παρόλα αυτά, τις καλύτερε ευχέ μου προ του Ρουμάνου συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Επίτροπο και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει να ανταλλάξουμε απόψεις για τα τόσο σημαντικά ε, αυτά θέματα. Για την ενιαία αγορά συγκεκριμένα που είναι από τους πυλώνες της Ένωσης. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί φραγμοί ωστόσο και δεν κάνουμε αρκετά, αρκετά σύντομα για να τους ε, αντιμετωπίσουμε. Παρόλα αυτά, σας ευχαριστώ για μια πολύ αναλυτική παρουσίαση. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα περιοριστώ στα εξή. Πρώτον, ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών που είναι ακρογωνιαίος λήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ συχνά ότι οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα εάν θέλουν να δραστηριοποιηθούν εκτός των συνόρων της χώρας ε, όπου εδρεύουν. Θυμάμαι ότι ενεκρίθη μια οδηγία κατά την τσεχική προεδρία για την κοινή αγορά υπηρεσιών. Οπότε η ερώτησή μου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα στον τομέα αυτό. Γιατί πολλοί από τους φραγμούς είναι συχνά απλώς ε, γραφειοκρατικής φύσης. Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Τι θα κάνετε για να τους αντιμετωπίσετε περαιτέρω Και κάτι άλλο. για την ε, διανοητική ιδιοκτησία, τα πνευματικά δικαιώματα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει μια ενιαία αγορά εδώ που παρέχει συμπληρωματική προστασία στα γενώσιμα φάρμακα για παράδειγμα. Χαίρομαι που περιλήφθηκαν όλα αυτά. Ξέρω ότι είναι ένα ειδικό τμήμα της αγοράς πολύ ιδιαίτερο και προβλέπεται μία εξαίρεση για τις εισαγωγές τρίτων χωρών. Αν δεν αντιμετωπιστεί όμως αυτή η εξαίρεση ε, σε το χρονικό διάστημα, τότε πολλά από αυτά τα γενώσιμα δεν θα μπορούν να παραχθούν πλέον στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει γιατί είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι που είστε μαζί μας σήμερα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπιούρκ. Ευχαριστώ για όλες ε, αυτές τις πληροφορίες ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Ε, η ανταγωνιστικότητα είναι πολύ σημαντικό για όλους στην Επιτροπή μας. Όλοι χρειαζόμαστε ένα σαφές νομικό πλαίσιο που να στηρίζει τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πολλά εμπόδια σε αυτό το τομέα και γι' αυτό οι επιχειρήσεις μας ε, δεν επιτυγχάνουν ε, στις διεθνείς αγορές το επίπεδο ανταγωνιστικότητας που θα ήθελαν. Οπότε θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπε και ο προηγούμενος ε, ομιλητής, τα γενώσιμα. Η πρόσβαση των επιχειρήσεών μας ε, στις αγορές των τρίτων χωρών είναι περιορισμένη. Διότι στις άλλες χώρες οι οι επιχειρήσεις μπορούν να ξεκινήσουν την παραγωγή αυτών των γενοσύμων πολύ νωρίτερα από ό,τι οι δικές μας επιχειρήσεις. Γιατί υπάρχουν ε, πολλές πιστοποίησεις που πρέπει να λάβουν οι δικές μας επιχειρήσεις. Υπάρχουν κανόνες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις εξαγωγές μας ε, γενοσύμων στις τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι αυτή η προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν είναι ευέλτιστη. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και αν βελτιώσουμε εδώ λίγο την κατάσταση, τότε θα δημιουργούσαμε και θέσει εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ. Ένα μόνο σχόλιο. Στην στρατηγική της ενίσχυσης της ιενές αγοράς, ένα τμήμα ασχολείται με τη συνεργατική οικονομία που περιλαμβάνει πολλούς επένους όπου τονίζει τις αρετές αυτών των νέων προτύπων και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Ωστόσο, πρέπει να τονίσω ότι υπάρχουν ε, πολλά πλεονεκτήματα γενικότερα για την διαφοροποίηση της παραγωγής προϊόντων και για τη μείωση του κόστους. Όμως δεν αναφέρονται καθόλου οι κίνδυνοι, ούτε μια γραμμή για την επίπτωση αυτών των νέων τύπου επιχειρήσεων και εμπορίου και για τις ε, ανησυχίες ε, για τα προβλήματα του ρυθμιστικού πλαισίου. Η μεγαλύτερη πρόκληση που θέτει η συνεργατική οικονομία πέρα από την αναγκαιότητα ενίσχυσης ε, των εγγύσεων προς τον καταναλωτή είναι στον τομέα της προστασίας των εργαζομένων. Σίγουρα η συνεργατική οικονομία σε ορισμένες περιπτώσεις επιτρέπει περισσότερη ευελιξία και συνδυασμό εργασίας και οικογενειακού βίου αλλά βλέπουμε ότι αυξάνεται επίση η επισφάλεια και μειώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων. Κυρία Επιτροπέ, ειλικρινά, πρέπει να υπάρξει περισσότερη πρωτοβουλία της Επιτροπής και αντιμετώπιση του κλάδου αυτού. Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, εδώ είμαι, από την άλλη μεριά. Εδώ, κοιτάξτε με, εδώ είμαι. Εδώ, εδώ, εδώ. Ωραία, τόσο το καλύτερο. Πρώτον, αυτό και τη βιομηχανία εκπομπές. Η πρόταση της Κομισιόν, όπως μας την παρουσιάσατε, είναι θαυμάσια. Υπάρχουν θέματα που είναι σχεδόν ανέφικτα. Αλλά πρέπει να τα επιχειρήσουμε παρόλα αυτά λόγω των όσων έχουν συμβεί. Σας παρακαλώ ποια είναι η εκτίμησή σας, τι θα σήμαινε αν εμείς ως Κοινοβούλιο στείλουμε πίσω το θέμα αυτό. Τι επιπτώσεις ε, θα είχε για την αυτοκινοβιομηχανία Να τονίσω ότι στην Ευρώπη ε, απασχολεί ο κλάδος αυτός 12 εκατομμύρια εργαζόμενους. Σκεφτείτε πώς είναι ένα αυτοκίνητο. 75% της προστιθέμενης αξίας του οχήματος προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζόμενους. 75 μικρομεσαίες. Από μικρομεσαίες. Εάν συνεχώς οξύνουμε τις προδιαγραφές, τι θα επιτύχουμε. Ξέρουμε ότι υπήρξαν ε, εγκληματικές ενέργειες μια συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν πρέπει να φυγεί ολόκληρος ο κλάδος. Δεύτερο θέμα. Ε, πυροβόλα όπλα για κυνήγι στα πλαίσια της οδηγίας για τα πυροβόλα όπλα. Όπως ξέρετε, πολλοί ε, κυνηγοί ανησυχούν, πολλοί που ε, αθλούνται στη σκοποβολή ανησυχούν για το μέλλον τους και μας βομβαρδίζουν με μηνύματα. Φαίνεται ότι αυτοί οι κυνηγοί και αυτοί οι αθλητές κοποβολής ε, εξομοιώνονται με τους ε, τρομοκράτες. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα. Κυκλοφορούν πολλές ε, φήμες για το τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν. Μήπως θα μπορούσατε και εδώ να διευκρινίσετε κάπως την κατάσταση για να μην συμβούν τα χειρότερα που πολλοί φοβούνται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είναι πολύ κοντά στα θέματα της ζωική ευζοίας η ερώτησή σας. Ο κύριος Γκίρεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να μιλήσω για την αυτοκινητομηχανία στην Ευρώπη, που δεν είναι μια ομοιόμορφη αγορά. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία, η Ρουμανία με μεγάλες αποκλήσεις. Και αρκετές άλλες. Ο μέσος όρος ζωής των ε, αυτοκινήτων είναι 13 χρόνια λόγω χάρη στην Πολωνία. Και αυτό έχει να κάνει και με πολύ μεγάλες ποσότητες εκπομπών, κυρίως αζωτούχων. Θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθούμε με αυτό σε επίπεδο μικρομεσαίων. Δεν μπορούμε να έχουμε ομοιόμορφη δράση σε όλη την Ευρώπη, διότι δεν υπάρχουν οι ανάλογες νομοθετικές ρήτρες. Ιδίω όπου έχουμε να κάνουμε με μονοπόλια στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Υπάρχει λοιπόν εδώ ένα σοβαρό σφάλμα που θα μπορούσε ενδεχομένως να διορθωθεί εάν η ρήτρα διόρθωσης ενεκρινόταν ε, από όλα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα αποτελέσουμε τροχοπέδι για την ανάπτυξη της, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αυτή την περίπτωση και θα μπορούμε ταυτόχρονα να ελέγξουμε και τις εκπομπές αριών του θερμοκηπίου με αυτή τη ρήτα της διόρθωσης, ε, το retrofit δηλαδή, την επισκευή, θα μπορούμε να επιφέρουμε τις ανάλογες ε, διορθώσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ζούμπιχ. Ευχαριστώ ε, Επίτροπε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σκληρή σας δουλειά και την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι πρωτοβουλίε για την επιχειρηματικότητα είναι πραγματικά επιτυχημένε και θα ήταν ιδιαίτερη χαρά μα να μπορέσουν να παραταθούν. Χθε μόλι συζητήσαμε την ιδέα των ε, γυναικών επιχειρηματιών, των business angels. Ε, υπάρχουν ε, μάλιστα τέτοια θέματα πολύ σοβαρά σε πολλέ χώρε τη Ευρώπη, με σοβαρά ποσοστά γυναικεία αδερφία. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε με τέτοια ενθαρρυντικά βήματα και να δούμε τι μπορεί να γίνει και για την μικροεπιχειρηματικότητα. Ε, βλέπουμε ότι ένα εκατομμύριο πρόσφυγες έχουν ήδη περάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως να είναι διπλάσιος ο ρυθμός του χρόνου. Δεν ξέρω λοιπόν κατά πόσον θα μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην αγορά εργασίας, αλλά σίγουρα κάποιο είδους απασχόληση πρέπει να βρεθεί και για αυτούς. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να ωφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές. Η επιχειρηματικότητα είναι ό,τι πιο σκόπιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Μόνον έτσι θα βρούμε κοινέ προσεγγίσεις και θα μπορέσουν οι προδιαγραφές μας να αναβαθμιστούν. Ο στόχος να έχουμε 20% περισσότερη παραγωγή στην Ευρώπη ως το 2020 είναι αξιέπαινος, αλλά προκειμένου να τον πετύχουμε θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι. Για την ώρα καθυστερούμε, χωρούμε. διότι ωραία θα ήταν να μπορούμε να υποσχεθούμε 30% περισσότερη παραγωγή στην Ευρώπη στο 2030, αλλά θα πρέπει να προλιάνουμε το έδαφο για κάτι τέτοιο. Και αυτό που χρειάζεται να προβλέψουμε είναι τι θα γίνει με την ε, κοινωνική πρόνοια και τι καλέ θέσει εργασία για όλου. Δηλαδή, όχι να γίνει κοινό αγαθό η φτώχεια ω προ την ενεργεια θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, είναι ακρογωνίως λίθος για να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τα βλέπουμε όλα ως αρνητικά. Ευχαριστούμε κυρία Μόντ, Ε, Ευχαριστώ να συμπληρώσω τα σχόλια του συναδέλφου Μπλάνκο Λόπες για την συνεργατική οικονομία, την συμμετοχική οικονομία και να μην ξεχνάμε την ομάδα ζωτικής σημασίας των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό το τομέα. Κατά δεύτερον, καλωσορίζω το γεγονό ότι αναφέρατε την κυκλική οικονομία για να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα με την κυκλική οικονομία θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ε, ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Όχι απλώς ε, επισκευές αλλά πραγματικά όλο το φάσμα των πολιτικών μας αποφάσεων. Αναμένω λοιπόν διακάω τι προτάσεις σας και ελπίζω να είναι φιλόδοξες, θα τις δούμε αύριο. Τρίτον, μιλήσατε για το διάστημα. Ένας τεράστιος κλάδος ως προς τη σημασία του και τους τομείς που καλύπτει. Είτε τις κλιματικές αλλαγές, είτε την άμυνα, την ασφάλεια, ακόμη και την υγεία ή άλλους τομείς. Νομίζω πάντως ότι έχουμε ακούσει να έχει προκληθεί σύγχυση σε αυτόν τον κλάδο ε, ως προς το που προσφέρονται διαφορετικές δυνατότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού για το διάστημα. Ε, καλωσορίζω τις απόψεις σας. Ελπίζουμε να έχουμε μια εικόνα του τι ε, θα προσφέρει η διαστημική στρατηγική για να ξεφύγουμε από κάποια από αυτά τα διέξοδα. Επίση, ελπίζω να υπάρχει περισσότερη ευλογία και του Κοινοβουλίου στα θέματα του διαστήματο, διότι για την ώρα σε αυτό το σημείο οι σχέσεις μας σημαδεύονται από κενό. Καλό θα ήταν να υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και για αυτή την κατεύθυνση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Βερκούναν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γιορτάζουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας μας την Κυριακή. Ίσως λοιπόν να μιλήσω και εγώ φυναδικά καλύτερα. Θα τα προτιμήσω. Ε, ευχαριστούμε, Επίτροπε. Ευχαριστούμε για την ε, παρουσίασή σας. Έχω και εγώ μια σειρά από ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να στηρίξω όσα είπαν οι συνάδελφοι για την ε, συμμετοχική οικονομία είναι μέρος του προγράμματος για την επόμενη χρονιά και ξέρουμε ότι υπάρχει μια σειρά από εταιρείε στην Ευρώπη που έχουν αντιμετωπίσει δυσκολίες διότι το νομοθετικό πλαίσιο, είτε το εθνικό είτε το ευρωπαϊκό, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξή τους. Τις, θεωρεί κάτι σαν είναι όπως το παράδειγμα της ε, Airbnb. Σε μερικές χώρες αυτό ακόμα και μπορεί να απαγορεύεται. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε εάν για ίδιες υπηρεσίες μπορούμε να ορίσουμε παρόμοιους ρόλους. Η Airbnb δεν είναι ξενοδοχείο, ε, ούτε μπορεί να έχει ανάλογους φόρους. Θα πρέπει αυτά λοιπόν να φροντίσουμε να τα ρυθμίσουμε, να ευθυγραμμιστεί η λειτουργία τέτοιων εταιριών. Η μεικτή οικονομία λοιπόν, η συμμετοχική οικονομία είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα θέλαμε να το προχωρήσετε. Το δεύτερο θέμα είναι το μέλλον της ενιαίας αγοράς. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στη σημασία της ε, ενιαίας αγοράς, ιδίως με την κρίση των προσφύγων σε εξέλιξη. Ήδη άρχισαν οι έλεγχοι στα σύνορα σε κάποιες χώρες, μην το ξεχνάμε. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ε, πολιτών είναι βεβαίως ζωτική σημασία για μας, αλλά θα πρέπει να, σκεφτούμε και το τι ε, επιπτώσεις θα έχουν οι νέοι έλεγχοι στα σύνορα για την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να την προστατεύσουμε την εσωτερική αγορά. Και να σταθώ σε ένα σημείο που ανέφερε ο Μάρκος Πίπερ. Ε, μας απασχολεί η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα και στη χώρα μας. Έχουμε την δυνατότητα οπλοφορίας σε κάποιες περιπτώσεις ε, για δασοφύλακε στη χώρα μας, αλλά με βάση αυτή την οδηγία θα απαγορευτεί η χρήση τους. Θα θέλαμε λοιπόν να μπορέσουμε να προβλέψουμε κάποια εξαίρεση για αυτές τις περιπτώσεις στη Φιλανδία τουλάχιστον, ως συνάδελφος με αυτά. Με συγχωρείτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Σας εύχομαι και εγώ. Ε, ό,τι καλύτερο για την επέτειο του ρουμανικού λαού, αλλά να θυμίσω ότι το ίδιο και για την ε, χαλιβουργία στη Γαλλία είναι μια επέτειος για μας. Νομίζω δεν μπορούμε να μιλάμε για την εσωτερική αγορά χωρίς να αναφέρουμε τον ε, υπόλοιπο κόσμο. Με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για την ενιαία αγορά χωρίς να μιλούμε για τον ε, υπόλοιπο κόσμο διότι ό,τι προσπάθεια και να κάνουμε στην ανταγωνιστικότητα για να στρίξουμε τον κλάδο μας, αυτό προσπαθούμε τουλάχιστον, ε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα αν κάποιοι χρησιμοποιούν εργαλεία που αντίκενται στους κοινού μας κανόνες. Με ένα απλό κλικ θα μπορέσουν να πλήξουν την ανταγωνιστικότητά μας και θα έχετε καταλάβει τι εννοώ. Εννοώ την εταιρική σχέση που έχουμε ή που επιθυμούμε να αποκτήσουμε με την Κίνα. Ε, Όντω, η Κίνα δεν έχει καθόλου του ίδιου κανόνε με εμά και ο κόσμο ε, ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τη βιομηχανία ανησυχεί πάρα πολύ για την ε, εξέλιξη των σχέσεων με τη χώρα αυτή. Θα δυσκολευτούν οι δικέ μα επιχειρήσει και η πολιτική διαχείριση του νομισματό τη, του Γιάνν, είναι κάτι που και το χρησιμοποιούν προ όφελό του και το διαχειρίζονται όπω θέλουν. Μπορεί λοιπόν αυτό να ε, είναι αρνητικό για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Στην ενιαία αγορά λοιπόν θέλουμε κοινού κανόνε για να μην υπάρχει νοθεμένο και αθέμητο ανταγωνισμό. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο εκείνα λοιπόν. Υπάρχει και η κρίση του, χάλι, του τσαλιού. Ένα θέμα που το παρακολουθείτε στενά θα είναι πολύ ε, δύσκολο να βρούμε τα όπλα που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και έπειτα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τα διπλώματα ευρεσιτεχνία και με την ε, τεχνογνωσία. Οποιαδήποτε εταιρεία θέλει μπορεί να μετακινηθεί στην Κίνα, αλλά έχουν την υποχρέωση να έχουν joint venture με, την, κάποια κινέζικη επιχείρηση. Αναγκάζονται να μοιραστούν λοιπόν και τα διπλώματά μα και την τεχνογνωσία μα. Αυτό θα είναι λοιπόν Κάτι που μπορεί επίση να μα δημιουργήσει προβλήματα. Και τρίτον, δεν ξέρω αν είναι ακριβώ το θέμα του χαρτοφυλακίου σα, αλλά ω Επίτροπο μπορείτε να πάρετε θέση, πώ μπορεί η Ευρώπη να ε, προκαλέσει την δημιουργία και άλλων Ευρωπαίων πρωταθλητών σε στρατηγικού στρατηγικούς τομείς. Νομίζω ήρθε η στιγμή η Ευρώπη να προσδιορίσει ποια είναι η σκοπιμότερη γεωγραφική της αγορά. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε σε κάποιους τομείς ε, εξαγορές και συνενώσεις εκεί που υπάρχουν δεσπόζωσες θέσεις ενώ για κάποια άλλα προϊόντα που ακριβώ προέρχονται από την Κίνα και έχουν κατακλείσει την ε, διεθνή αγορά να σας θυμίσω ότι έχουμε το πρόσφατο παράδειγμα της Ιταλίας με την Group που ε, φέρνει ε, ανοξίδωτο ατσάλι σοριδών από την Κίνα και η Κίνα αυτή τη στιγμή κατέχει τουλάχιστον το 50% της παγκόσμιας αγοράς στα προϊόντα αυτά. Δεν ξεπεράσατε τα τρία λεπτά τουλάχιστον. <coughs> Για να μην πω δύο. Ο συνάδελφος Χέλμερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους πρέπει να πω ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι μέρα ανεξαρτησία σήμερα. Ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε μετά από το δημοψήφισμά μας να γιορτάσουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας μας. Να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την ενδιαφέρουσα ε, συζήτηση. Ε, το θέμα της ανταγωνιστικότητας ε, από τότε που έχουμε επαφέ μαζί σας έχει τεθεί πολλές φορές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, συμμερίζετε τη δική μου ανησυχία ότι οι ενεργειακές τιμές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών. Μήπως μπορώ να σας ρωτήσω κατά πόσο θα συζητήσετε με τους συναδέλφους σας στο Σώμα των Επιτρόπων που ασχολούνται με το θέμα της κλιματικής αλλαγής, ώστε να τους παροτρύνετε να αλλάξουν τις υπάρχουσες πολιτικές για να υπάρξει μια ε, προσβάσιμη και ασφαλής ενέργεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας ρωτήσω επίσης αν έχετε λάβει υπόψη ε, ε, τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων Έχουμε το θέμα αυτό που μας απασχολεί, αλλά με απασχολεί και το θέμα της διαρροής του άνθρακα. Κάνουμε ιδιαίτερη μνήα ε, στους εντατικούς χρήστες ενέργειας, όμως μήπως το σύστημα ETS δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες εσείς έχετε ιδιαίτερη ευθύνη. Ευχαριστώ πολύ πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, γιατί ε, δεν χρειαζόμαστε εμείς ε, ένα δημοψήφισμα για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε την ημέρα της ανεξαρτησίας σε όλες τις ε, χώρες μέλη. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, με συγχωρείτε που καθυστέρησα και δεν άκουσα την εισαγωγική σας παρουσίαση, αλλά διάβασα την στρατηγική σας για την ιστορική αγορά και θα ήθελα να αναφερθώ στα εξή. Πρώτον, η στρατηγική σας αυτή για τα ελεύθερα επαγγέλματα, γιατροί, οδοντίατροι, φορολογικοί σύμβουλοι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί. Δεν ξέρω αν το ανέφερε κανείς. Αυτές οι επαγγελματικές ομάδες που στη Γερμανία αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν δικές τους ε, οργανωτικές δομές. Βλέπω ότι θέλετε να τις καταργήσετε εμείς έχουμε επιμελητήρια για αυτά τα ελεύθερα επαγγέλματα στις χώρες μας που ε, διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο οργάνωσης και υψηλές προδιαγραφές και για την ε, κατάρτιση των επαγγελματιών. Και έτσι διευκολύνουν και το κράτος και τις κρατικές υπηρεσίες. Αυτές τις επαγγελματικές ενώσεις και τις ενώσεις όπου πρέπει να ε, πληρώνει κανείς για να συμμετάσχει, αυτές οι ενώσεις δεν είναι φραγμοί για την οικονομία διευκολύνουν το κράτος. Οπότε σας παρακαλώ να μην τις ε, παρεμποδίζετε. Ορισμένοι αναφέρθηκαν ήδη στο σκάνδαλο της Volkswagen. Τον υποστηρίζω, το είπε και ο Σάλφος Ρούμπιχ. Σας παρακαλώ βεβαίως να διελευκάνετε το σκάνδαλο. Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό. Αλλά να μην καταργήσετε την τεχνολογία diesel η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον Σας παρακαλώ ως αρμόδια για την ενιαία αγορά να φροντίσετε να υποστηριχθεί περαιτέρω αυτός ο κλάδος. Και τελευταίο σημείο, τα όπλα. Αναφέρθηκε ήδη. Και θέλω και εγώ να το τονίσω. Στη Γερμανία ε, είναι πολύ αυστηρός ο νόμος γι' αυτό. Πριν από κάποια χρόνια υπήρξαν κάποιες ε, περιπτώσεις εγκλημάτων και οξύναμε. Κάναμε ακόμη πιο αυστηρούς τους νόμους. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τώρα γιατί μέσω ευρωπαϊκής εναρμόνισης ε, επιδιώκεται υπεραιτέρω ε, προσπάθεια αυστηροποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάνκα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η εκβιομηχάνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι γεγονός ε, όμως ότι η βιομηχανική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μειωθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Έχω την εξής ερώτηση. Έχετε προσέξει ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ ενός ευρώ που είναι πολύ ισχυρό για τις, νότιες, για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης που δεν μπορούν να εξάγουν όπως έκαναν στο παρελθόν και από την άλλη ενός ευρώ που είναι πάρα πολύ αδύναμο για ε, ε, χώρες όπως η δική μου, η Γερμανία, όπου η εκβιομηχάνηση όλο και αυξάνεται. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Συμφωνείτε ότι υπάρχει ε, μια σχέση μεταξύ ενός ε, ενιαίου νομίσματος το οποίο πλήττει το νότιο τμήμα της Ευρώπης ε, και αποτελεί κάποιο είδους επιδότηση για, την, για το βόρειο τμήμα της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Όχι. Πολλές ερωτήσεις σας ε, απευθύνθηκαν, ε, κυρία Επίτροπε. Πάρα πολύ μας ενδιαφέρουν οι απαντήσεις σας, γιατί εκτός από τέσσερα θέματα, εκτός από τα τέσσερα θέματα, υπήρξαν και άλλα θέματα που ετέθησαν ε, εσωτερική αγορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανταγωνιστικότητα, διαστημική πολιτική. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. θα προσπαθήσω κάπως ε, οργανωμένα να απαντήσω στα ερωτήματα. Τα έχω σημειώσει όλα. Και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας με τη σειρά. Πρώτον, όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, γιατί πολύ θέσατε το σχετικό θέμα, Θέλω να το πω κατηγορηματικά αυτό. Δεν θέλουμε να ξεφορτωθούμε του κινητήρε δίζελ. Θέλουμε να ενισχύσουμε την αυτοκινητοβιομηχανία μα γενικότερα. Αυτό είναι απάντηση προ όλου εσά που κάνατε σχετική ερώτηση. Εγώ είμαι εδώ να σα παρουσιάσω την, ε, την βιομηχανική άποψη των πραγμάτων. Βέβαια πρέπει να λάβω υπόψη όλε τι συμφωνίε, τις δεσμεύσει μα, τι δεσμεύσει του Συμβουλίου και των, των κρατών μελών κατά τη διάρκεια και των προηγούμενων ετών. Η αυτοκινητοβιομηχανία πάντως ε, είναι πραγματικά ένα κόσμημα μεταξύ των τομέων μας. Πρέπει να το προστατεύσουμε, αλλά δεν πρέπει να κλείνουμε και τα μάτια σε περιπτώσεις απάτης όπως ε, συνέβη στην ε, περίπτωση αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι η καλύτερη απάντηση για την ώρα, στην κατάσταση στην οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, είναι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Οι καταναλωτές, γιατί άμα δούμε τα οικονομικά αποτελέσματα αυτού και του επόμενου ε, οικονομικού έτους, θα μας δείξουν ε, την αντίδραση των καταναλωτών ε, στην υπόθεση Volkswagen. Πρέπει να ανακτήσουμε, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τους και για να γίνει αυτό, δύο πράγματα πρέπει να συμβούν. Πρώτον, να υπάρχει ένας κύκλος δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες, σε πραγματικό χρόνο, είναι ένα γνήσιος, ένας γνήσιος τρόπος ε, να το κάνουμε αυτό και μπορούμε από το Σεπτέμβριο του 2016 με μια προοπτική 2 με τέσσερα έτη ε, να έχουμε πολύ πιο καθαρούς κινητήρες diesel. Αυτή είναι η προοπτική μας Μπορεί να έχουμε μια άλλη προοπτική για τα επόμενα 20-30 χρόνια, όμως πρέπει να, έχουμε, να, να αναλάβουμε να, να λάβουμε σιγά σιγά κάποια μέτρα και να πάμε ένα-ένα στα βήματα. Ο κύκλος δοκιμών σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι φιλόδοξο από τη μία ε, και είναι και πολύ καλό για το περιβάλλον γιατί θα μειώσει... ε, ε κατά το 1 τέταρτο ε, τις, ε, τις ε, εκπομπές είναι κάτι το οποίο αν δεν το κάνουμε δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Είναι κάτι στο οποίο η βιομηχανία ρίχνει πάρα πολύ χρήμα και δαπανά και πάρα πολύ ενέργεια. Είναι, ε, πρέπει, πρέπει να διατηρήσουμε τον σύγχρονο χαρακτήρα της αυτοκινητοβιομηχανίας μας, αλλά από την άλλη πρέπει και να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών που επλήγει όλος ιδιαίτερος. Και κάτι ακόμη το οποίο το συζητούσα την περασμένη εβδομάδα με τον εκτελεστικό διευθυντή της Volkswagen στο Στρασβούργο και του είπα και θα σας το πω και εσάς κατηγορηματικότατα ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξή κατάσταση, οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ να την χάνουν διαφορετική συμπεριφορά από του Αμερικανού. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει το περιβάλλον, υπάρχουν κάποιε οικονομικέ συγκυρίε διαφορετικέ ε, στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά η απάτη ήταν ίδια και εδώ και εκεί. Πρέπει να έχουμε το ίδιο επίπεδο αποζημίωση λοιπόν. Δεν ξέρω πώ ακριβώ θα επιληθεί αυτό το ζήτημα, αλλά μετά τη συνάντησή μου με τον εκτελεστικό διευθυντή υπήρξε μια δημόσια ανακοίνηση ότι δεν θα, γίνει, δεν θα υπάρξει αποζημίωση προς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από τη Volkswagen. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι παράδεκτο. Κύριε Νίκα, να σας ζητήσω συγγνώμη για την μακροχρόνια διαδικασία Είπατε ότι δεν σας έχουμε δώσει απαντήσεις. Ε, πράγματι είναι απαράδεκτο αυτό. Ακόμη όμως ε, προσπαθούμε στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης να αναπτύξουμε τις ε, ε, ικανότητές μας. Πράγματι συμμετέχω πάρα πολύ και είναι δική μου ευθύνη η ενεργειακή αγορά και ε, οι ενεργειακές τιμές γιατί είναι τμήμα του κόστου της βιομηχανίας. δεν είναι δυνατόν να υπεκφύγω, ούτε θέλω να το κάνω. Οπότε θα ήθελα να πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η Ενεργειακή Ένωση. Εγώ όμως απλώς παρουσιάζω τη βιομηχανική θεώρηση των πραγμάτων. Όσον αφορά τη, τα πιο μακρόχρονα ε, συμβόλαια ε, ενέργειας, πράγματι είναι καλύτερα από απόψεως σχεδιασμού. Εμείς παρακολουθούμε το ζήτημα και παρακολουθούμε και τις τιμές της ενέργειας. Σε μερικές περιπτώσεις και πρέπει να το πω και προς τον κύριο Χέλμερ, για τις ενεργειακές τιμές, για το χάλιβα, Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι θέμα ευρωπαϊκής νομοθεσίας, είναι θέμα εθνικής φορολογίας ε, που είναι πάρα πολύ υψηλή. Εγώ να το παρακολουθήσω το θέμα, γιατί τώρα συστήσαμε μια ομάδα που θα προσπαθήσει να δώσει όλες τις πληροφορίες για τις ε, πολύ υψηλέ ενεργειακές τιμές στα διάφορα κράτη-μέλη, αλλά σε μερικές περιπτώσεις ο λόγος δεν είναι κλιματική πολιτική, δεν είναι ε, ενωσιακή ε, ενεργειακή πολιτική, αλλά είναι θέμα εσωτερικής πολιτικής του κράτους μέλους. Και αυτή είναι η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου και πραγματικά πρέπει να το τονίσω αυτό. Όσον αφορά τα ε, γενώσιμα, επειδή δύο ευρωβουλευτές έθεσαν το ερώτημα αυτό, και μιλάω τώρα για τη συμπλήρωση των ε, πιστοποιητικών προστασίας και της ευρεσιτεχνίας. Εγώ έρχομαι σε επαφή με τη φαρμακοβιομηχανία και με τις εταιρείες γενοσύμων φαρμάκων. Θέλουμε να προγραμματίξουμε μια απαλλαγή κατασκευής ε, που θα δώσει τη δυνατότητα στη φαρμακοβιομηχανία να κατασκευάσει πάρα πολλά ε, γενώσιμα φάρμακα, αλλά επίσης να δώσει και πάρα πολύ ψηλού επίπεδου θέσεις απασχόλησης. Είναι κάτι το οποίο θα αναφέρεται στη στρατηγική μας για το επόμενο έτος και στο πρόγραμμα εργασίας μας ε, και στο πρόγραμμα εφαρμογής της στρατηγικής μας όσον αφορά τη συνεργατική οικονομία. Γνωρίζετε όλοι και το ανέφερα, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη σε σχέση με την προσέγγιση της ε, συνεργατικής οικονομίας. Εγώ προσωπικά πιστεύω, ίσως θα έπρεπε και εσείς να το λάβετε υπόψη στις συζητήσεις σας, ε, δεν είναι δυνατόν να καταπολεμήσουμε αυτό το νέο μοντέλο επιχείρησης, γιατί είναι άχρηστο, δεν πρόκειται να κερδίσουμε ποτέ αυτόν τον αγώνα όλο και περισσότερα ε, και καινούργιες εφαρμογές ε, εμφανίζονται και θα δημιουργήσουν ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με τρόπο ομοιογενή σε ολόκληρη την Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς είπα ότι με τις κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να εξασφαλίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αυτές ε, οι επιχειρήσεις πληρώνουν τους φόρους τους, ότι είναι δίκαιες προς τον εθνικό προϋπολογισμό και επίσης εφαρμογή. Εγώ δεν θα ήθελα να υπάρξει νέος κανονισμός. Θα υπάρξουν κατευθυντήριες αρχές, για, ε, κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία και του χαρτοφυλίου της Επιτρόπου Γιούροβα πώς ισχύουν για την συνεργατική οικονομία και θα ελπίσουμε να υπάρξουν ε, μέτρα ήπιας νομοθεσίας ε, στα κράτη-μέλη όσον αφορά την κυκλική οικονομία γιατί αυτό συνδέεται άμεσα με το θέμα των σωστών τεχνικών ελέγχων και της ε, επισκευής των ε, αυτοκινήτων. Ε, στην οδηγία για την έγκριση τύπου θα το καλύψουμε. Το πρώτο θέμα είναι η επιβολή της νομοθεσίας και το δεύτερο είναι η επιλογή της πιο ευνοϊκής νομοθεσίας, το, το shopping forum θα επικεντρωθούμε περισσότερο στη διαφοροποίηση των κρίσιμων πρώτων υλών, των ε, πόρων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, ε, το, ε, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των, ανανεώσιμων προϊόντων που μπορούν να ανακυκλωθούν. Είναι όμως ένα ζήτημα ε, το οποίο καλύπτει και η βιομηχανία αλλά και το περιβάλλον. Γιατί νομίζω ότι μόνο αν συμμετέχει και η βιομηχανία στην όλη διαδικασία ε, τα ανακυκλώσιμα και η κυκλική οικονομία θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε όλους μας τους στόχους που βεβαίως έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πακέτο. Όμως πρέπει η βιομηχανία να είναι φίλος μας ε, και όχι εχθρός μας. για κάποιες ε, ερωτήσεις ε, που αφορούν την οδηγία για τα ε, πυροβόλα όπλα. Κυνηγοί, ερασιτέχνες και όλοι όσοι έχουν ένα, αυτό το ευγενές χόμπι. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, πρέπει να αντιδράσουμε σε μια δραματική κατάσταση και το κάναμε αυτό. Ο στόχο αυτού του πακέτου, γιατί πρόκειται για ένα πακέτο, κανονισμό και οδηγία, είναι να αντιμετωπίσουμε βασικά ζητήματα ασφαλεία. Πρώτον, τον εντοπισμό των όπλων. Πρέπει να γνωρίζουμε, σαφώ υπάρχει βέβαια και το λαθρεμπόριο, αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι ο ιδιοκτήτη του κάθε όπλου και πώ μετακινείται το όπλο αυτό εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, να υπάρξει ένας, ε, μια απενεργοποίηση σε, με, με, με, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε τι έγινε στο Σαρλί είδαμε τι έγινε στο τρένο ταχεία στο Ταλής, τα ε, ε, όπλα που χρησιμοποιήθηκαν ε, είχαν αγοραστεί παρανόμως στο ίντερνετ. Κάποια άλλα ε, θεωρούσαν ε, οι αρχές ότι δεν υπήρχαν, ε, ότι είχε γίνει αποπλισμός αλλά τελικά δεν είχε συμβεί αυτό. Οπότε, πρέπει να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάποιος κυνηγό, συλλέκτης θέλει να αγοράσει νομίμως ένα όπλο να μπορεί να το κάνει, αλλά μετά, αλλά, αλλά μετά από αδειοδότηση πολύ συγκεκριμένη. Μετά θα υπάρχει μια άδεια χρήση των όπλων αυτών, αλλά πρέπει να ξέρουμε σε περίπτωση αγοράς ενός νέου όπλου όλες τις συνθήκες. Και μιλάω για παράδειγμα για τη χρήση για παράδειγμα των, των Καλάσνικοφ, για ιδιωτική χρήση. Εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας. Όσον αφορά τη χαλιβουργία. Πρώτον, για το ETS, το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων. Το έχω ξαναπεί. Εγώ παρουσιάζω την βιομηχανική θεώρηση των πραγμάτων. Δεν μπορώ να συμφωνήσω Είναι γεγονός ε, αυτό που είπατε ότι το ETS έχει, κάποιο, έχει κάποια, εμ, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις που έχουμε λάβει δεν μπορούν να προχωρήσουν. Γιατί εμείς Δεν πρέπει να λάβουμε τις λάθος αποφάσεις που μπορεί να πλήξουν πολύ σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα την Κίνα. Είμαι σε ασθενή συνεργασία με την Επίτροπο Μάλμστρομ ως προς το θέμα αυτό και συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Μαρτά ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε εμπορικό μέσο έχουμε στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε ένα ισότιμο πεδίο για τη δική μας βιομηχανία, εμπροκειμένου στον τομέα της ε, χαλιβουργίας. Θα συζητήσουμε επίσης και το θέμα της ε, ε, ελεύθερης αγοράς με την Κίνα είναι πραγματικά ένας τεράστιος κίνδυνος για τη δική μας αγορά, όχι μόνο για τη χαλιβουργία και για άλλους τομείς. Αν είμαστε απολύτως ανοιχτοί και αν δώσουμε τέτοιου είδους καθεστώς στην Κίνα, νομίζω ότι πρέπει να γίνει κατόπιν συζήτηση ε, υπό διάφορε οπτικές γωνίες, μεταξύ των οποίων και τη βιομηχανική βεβαίω. όσον αφορά τα ελεύθερα επαγγέλματα. Να πω κάτι που το είπα και στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Έχουμε 5.000 ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ε, στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το είπατε και εσείς κυρία Νίμπλερ ε, πράγματα τα οποία έχουν πει ε, ε, ενώσεις τέτοιου είδους επαγγελμάτων στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο πάντοτε την ίδια επαναλαμβανόμενη επιχειρηματολογία ακούμε ότι αν απελευθερωθεί ένα επάγγελμα θα αποτελέσει κίνδυνο για την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών. Κοιτάξτε, δεν θα φτάσουμε ποτέ σε μια τέλεια κατάσταση. Και σαφώ υπάρχουν ευαισθησίε μεταξύ των κρατών μέλων, διαφορετικέ οικονομικέ συγκυρίε σε κάθε κράτο μέλο. Όμω, η βασική ιδέα πρέπει να επαναλαμβάνεται και να εφαρμόζεται. Ότι έχουμε πολύ περισσότερα ελεύθερα επαγγέλματα ε, στην Ευρώπη, γιατί βάση είναι η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και σε γενικές γραμμές δεν ισχύει ότι αν κάποιος ανήκει σε μια τέτοια ένωση ε, ελεύθερων επαγγελμάτων στην Ισπανία, το να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες αυτές είναι πιο επικίνδυνο από το να είναι κανείς μέλος σε μια ένωση μια άλλης χώρας μέλους. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχω επαναλάβει πολλές φορές τα 28 κρατη γιατί προστατεύουν τις δικές τους αγορές. Καταλαβαίνω βέβαια ότι υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά, αλλά θα πάμε γενικά προς την κατεύθυνση των φιλελεύθερων επαγγελμάτων. τη απελευθέρωση των επαγγελμάτων. Για το διάστημα και την διαχείριση του διαστήματος. Είναι λίγο νωρί να πω τι μορφή θα έχει η Ευρωπαϊκή Στρατηγική το διάστημα. Αλλά χθε ακόμη συζητούσαμε με την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου γιατί μετά από πολλά χρόνια, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει πολύ σοβαρά τις αρμοδιότητές της για τα θέματα του διαστήματος και τον κλάδο του διαστήματος. Η στρατηγική θα εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του Διαστήματος, Νορβηγία και Ελβετία επίσης θα συμμετάσχουν από τον ΝΕΟ γιατί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Μετροπή μάλλον, είναι το θεσμικό όργανο που κατεξοχήν χρηματοδοτεί σχεδόν κατά 100% της δράσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Διάστημα. Πρέπει να δεχτείτε την άποψή μας που είναι τελείως σαφής και δεν αμφισβητείτε. Θέλουμε να έχουμε και επιρροή και πολύ ξεχωριστό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών από τον οργανισμό. Αυτά ευχαριστώ. Thank you very, very much. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Πάρα πολλές ερωτήσεις, μακροσκελέστατη, διεξοδική και βαθιά συζήτηση. Τέτοιο διάλογο, διαρθρωμένο διάλογο, σε μηνιαία βάση ε, είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε. Γιατί τα βλέπουμε τα πράγματα από τη σκοπιά της νομοθεσίας, αλλά γνωρίζουμε και τη δική σας την οπτική γωνία, τις δραστηριότητές σας, τις αποφάσεις σας, τι κάνετε. Όλες οι ερωτήσεις είναι πολύ εύστοχες. Και αυτό βεβαίως σας δίνει και την ε, δυνατότητα να προετοιμάσετε τι μελλοντικέ σα δραστηριότητε, Επίτροπο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όλοι θα λάβετε γραπτέ απαντήσει στι ερωτήσει σα πολύ γρηγορότερα από ό,τι προηγουμένω. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ευχαριστούμε. Ευθύ αμέσω περνάμε. Uh, uh, thank you, colleagues. And let me apologize from the very, very beginning. Ευχαριστώ, ε, συνάδελφοι. Ευθύς αμέσως να ζητήσω συγγνώμη από την προσκεκλημένη, την επόμενη προσκεκλημένη της Επιτροπής μας, την κυρία Ντομενίκ Ριστόρη, η οποία περιμένει τουλάχιστον εδώ και 20 λεπτά. Ο κύριος Ντομενίκ Ριστόρη μάλλον. Ε, μας συγχωρείτε που σας κάναμε να περιμένετε, αλλά είναι μεγάλη μας χαρά που είστε εδώ μαζί μας και μπορούμε να έχουμε μια πλήρη και ενδελαχή συζήτηση για το θέμα της σας διάταξης. Δεύτερος κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος. Κύριε Γενική Διευθυντά, αγαπητέ Ντομινίκ, Εάν μπορείτε να πείτε λίγα πράγματα και για τον πρώτο κατάλογο, γιατί το να μιλήσουμε για τον δεύτερο κατάλογο χωρίς να γνωρίζουμε τον πρώτο, είναι λίγο αναρθόδοξο. Θα ήταν ωραίο λοιπόν να γνωρίζουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο καταλόγων. Αλλά εδώ μας απασχολεί ο δεύτερος κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος για τη σημερινή μας συζήτηση για την εσωτερική αγορά ενέργειας, για την ασφάλειά μας, για τα θέματα του κλίματος, όσα θέλουμε να πετύχουμε στο μέλλον. Και την Ενεργειακή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και έχετε το λόγο, κύριε Γενική Διευθυντά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, διότι οι υποδομές της ενέργειας διαδραματίζουν το ρόλο στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης. Εν είδη εισαγωγής θα ήθελα απλώς να κάνω τρεις παρατηρήσεις αυτής της εξορχής. Πρώτα απ' όλα η καλά διασυνδεδεμένη αγορά είναι η βάση για να έχουμε ολοκληρωμένη ανταγωνιστική και βιώσιμη εσωτερική αγορά ενέργειας γνωρίζω ότι και από σας προσωπικά και συλλογικά έχουμε τη στήριξή σας για την εσωτερική αγορά ενέργειας. Δεύτερον, πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι από τους, έχει ένα από τα πιο προηγμένα δίκτυα αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υποδομές τους. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο και ευθυνές. Όσες φορές συμμετέχω σε διεθνείς συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, λαμβάνουμε φιλοφρονήσεις και συγχαρητήρια ακόμη και από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές μας ή τους εταίρους μας, οι Πολιτείες λόγω χάρη, αναγνωρίζουν την έμπειρο γνωμοσύνη μας σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Δίκτυο γενικώς Τρίτον, ένας από τους βασικούς μας στόχους ήταν, όπως καλά γνωρίζετε, να πάυσει η λεγόμενη ενεργειακή απομόνωση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να σας ε, αναγγείλω ότι σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν έχουμε διαδραματίσει σημαντική πρόοδο. Σε δύο εβδομάδες θα πάω στη Λιθουανία, στο Βίλνιος, για να εγκαινιάσω δύο σημαντικές εσωτερικές διασυνδέσεις. Ε, το Λιτπολ, ε, Λιθουανία, Πολωνία και το Λιτμπάλτ, Λιθουανία, Βαλτική διότι η διασύνδεση Σουηδίας-Λιθουανίας και Πολωνίας-Λιθουανίας είναι σοβαρότατες προσθήκες με 200 ΜΒ ως προς το δυναμικό της διασύνδεσης και ένα νέο σύνδεσμο μεταξύ τελείως απομονωμένων χωρών κατά τα άλλα. Και με διασύνδεση και της υπόλοιπης Ευρώπης μεταξύ με, μέσω της Πολωνίας και της Σουηδίας. Ένα άλλο παράδειγμα, το περασμένο Φεβρουάριο, τα εγγένεια της νέας ηλεκτρικής γραμμής μέσα από τα Πυρηναία που συνδέει την Γαλλία με την Ιβερική Χερσόνησο, διπλασιάζοντας το επίπεδο διασύνδεσης μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Άλλη μια πρόσφατη επιτυχία μας, η υπογραφή πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου του κύπελ, ε, του νέου ε, αγωγού αερίου μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας, 400 χιλιόμετρα τουλάχιστον μεταξύ Πολωνίας και Βαλτικών χωρών. Πολύ σημαντικό από κάθε άποψη. Σε ό,τι αφορά το νέο κατάλογο των έργων κοινού ενδιαφέροντος, να πω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει 195 ε, μεγάλα έργα υποδομών. Η προετοιμασία μας ήταν πάρα πολύ καλή με συμμετοχή όλων των βασικών φορέων, όχι μόνο των μελών, ρυθμιστών, TSO, Ευρωπαϊκών Οργανισμών, κοινωνίες των Πολιτών και σε σύγκριση με τον πρώτο κατάλογο που είχε εγκριθεί το 2014 η διαφορά είναι η εξή. Ο νέος κατάλογος περιλαμβάνει 108 έργα ηλεκτρισμού. 77 για το φυσικό αέριο, 7 για το πετρέλαιο και 8 για τα εφή δίκτυα. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο κατάλογο, ο νέος κατάλογος έχει 52 λιγότερα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Ήδη τα περισσότερα έχουν ανατεθεί ή θα ανατεθούν επιτυχώς στο τέλος της χρονιάς και έχει μειωθεί ο ρυθμός έργων στον τομέα του αερίου ε, αντιμετωπίζοντας έτσι τα σημεία όπου υπήρχε συμφόρηση. Θα μπορέσουμε να εξορροπήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο καλύτερα την ηλεκτρική ενέργεια με το αέριο λόγω και των πολιτικών ε, στόχων του Κοινοβουλίου, των πολιτικών επιθυμιών του Κοινοβουλίου και την ε, μεταμόρφωση του ενεργειακού μας συστήματος. Επιπλέον, να πω λίγα λόγια και για τη μεθοδολογία μας. Επικεντρωθήκαμε στα εξής σημεία πρώτα απ' όλα τα, τα δεκαετή προγράμματα ανάπτυξη δικτύων. Μόνον έργα που μπορούν να ενταχθούν σε αυτά τα δεκαετή προγράμματα είναι ρέσμα για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος. Επίτα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη υποψηφιότητα, αλλά και το κριτήριο της περιφερειακής ομαδοποίησης για να αξιολογήσουμε και να βαθμολογήσουμε σωστά τα υποψήφια έργα. Κοιτάξαμε και την ποιοτική και την ποσοτική διάσταση, όπως ορίζονται στον κανονισμό. Και για πρώτη φορά τα έργα επιλέγονται βάσει της ε, ανάλυσης κόστους ωφελίας, της διεταυρώμενης ωφελίας, βάσει της μεθοδολογίας που έχει αναπτυχθεί από, τους NSO από το ένσο E και το nso G και η κοινωνία των πολιτών συμμετείχε. Είχαμε δημόσιες διαβουλεύσεις καθώς και ε, σοβαρότατες συνομιλίες με όλους τους ε, ενδιαφερομένους φορείς. Στηρίζουμε και νέες πρωτοβουλίες όπως την εταιρική σχέση για την πρωτοβουλία των εφείων δικτύων ε, συνδυάζοντας ταυτόχρονα και TSO και NGO ε, πρέπει να πω ότι ο περιφερειακός κατάλογος ε, ούτως ή άλλως εγκρίθηκε συνετικά, δηλαδή ομόφωνα. Τον στήριξαν όλα τα κρατημέλη, κάτι που είναι αξιοσημείωτο. Τη στιγμή πρέπει να φανούμε ενωμένοι για να στηρίξουμε τα σημαντικότερα προγράμματα ενέργειας και έργα ενέργειας. Ως προς τα ωφέλη που θα αποκομίσουμε από αυτά τα έργα, κοινού ενδιαφέροντο. Ας διαχωρίσουμε τον ηλεκτρισμό και το αέριο. Στον ηλεκτρισμό η έγκαιρη υλοποίηση των έργων σημαίνει ότι θα μπορέσουν 26 κράτη-μέλη να επιτύχουν το στόχο του 10% διασύνδεσης με ηλεκτρική ενέργεια στο 2020 που έχουμε θέσει. Η Κύπρος και η Ισπανία θα ακολουθήσουν με μια μικρή καθυστέρηση αλλά αυτό είναι σημαντικό γιατί ξέρω ότι στηρίζετε τη διασύνδεση του 10% και εσείς. Η αλληλοδιασύνδεση είναι ύψιστη ε, προτεραιότητα για να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρχει ε, εύρυθμη ροή ηλεκτρικής ενέργειας από το ένα σημείο τη Ευρώπη στο άλλο, από το βορρά στο νότο και από τα ανατολικά προς τα θετικά. Ε, επίσης, θα αντιμετωπίσουμε πολλά σημεία συμφόρησης ε, για την ενέργεια στη Γερμανία, το Βέλγιο, την ε, Ολλανδία, την Αυστρία και ούτω καθεξής. Στην Ανατολική και την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη νέοι διασυνδέτες μεταξύ Ουγγαρίας, Σλοβακίας, Γερμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας Όλα αυτά θα αυξήσουν τις δυνατότητες ε, μεταφοράς ενέργειας στην κάθε περιφέρεια. Στην Βαλτική ξέρουμε τη μεγάλη επιτυχία του Μπενί που ξεκινήσαμε και με τη δική σας στήριξη και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αντιμετωπίσουμε όλα τα σημεία συμφόρησης για να υπάρχει καλύτερη διασύνδεση αλλά και να αντιμετωπίσουμε την απόλυτη εξάρτηση κάποιων χωρών, ιδίω των Βαλτικών. το ίδιο και στην Βόρεια Θάλασσα. Διότι θα υπάρξουν νέοι διασυνδέτες που θα εξυπηρετήσουν κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ώστε να επιτύχουν το στόχο αλληλοδιασύνδεσης μέσω διαφορετικών έργων. Σε ό,τι αφορά το αέριο, έχουμε εντοπίσει έργα που θα συμβάλλουν στην διαφοροποίηση της ε, προμήθειας του εφοδιασμού. Τα hub που θέλουμε να δημιουργήσουμε κυρίως στον χώρο της Μεσογείου, τα κομπικά σημεία δηλαδή και η καλύτερη πρόσβαση στην ενέργεια είναι σημαντικά στοιχεία. Άκρος σημαντικό προκειμένου να ε, εφαρμόσουμε σωστά τη στρατηγική για την, ε, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης θα δώσουμε έμφαση στα προγράμματα, στα έργα κλειδιά για τις πιο ευάλωτες περιοχές. Στην Δυτική Ευρώπη το ΜΙΚΑ ε, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας θα διευκολύνει την μεταφορά αερίου από τα νότια προς τα βόρεια αλλά θα εξυπηρετήσει και την ενίσχυση των επιδόσεων της αγοράς αερίου τοπικών. Το ίδιο στην κεντρική, ανατολική και νότιο-ανατολική Ευρώπη. Με στρατηγικές εγκαταστάσεις ενέργειας στην Κροατία λόγου χάρη, την Ελλάδα, Η ε, διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, Βουλγαρίας-Ρουμανίας, Σλοβακίας-Ουγγαρίας θα βοηθήσουν την διαφοροποίηση του εφοδιασμού για τις πιο ευάλωτες περιοχές. Και αυτό θα μπορέσουμε να το επιδιώξουμε και στην περιοχή της Βαλτικής. Περίπου 60 έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2017. Τα έργα αυτά θα ωφεληθούν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από το ενισχυμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, που όπως ξέρετε έχουμε εμείς το πλεονέκτημα να έχουμε αναπτύξει ένα από τα πιο προηγμένα ρυθμιστικά πλαίσια στον κόσμο. Κάποιες φορές έχει τόσο καλέ επιδόσει στο αριθμητικό μα πλαίσιο που τελικά καταλήγει να γίνεται τροχοπέδι. Επίση θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και ευθυγράμμιση τη διοικητική ε, προσέγγιση. Και ολοκληρώνω λέγοντα ότι θα ε, αξιοποιήσουμε όλα μα τα μέσα και εργαλεία. Βεβαίω το. Ε, η διευκόλυνση για τη διασύνδεση τη Ευρώπη. Το ΕΦΣΙ, το, το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, είναι εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να οδεύσουμε ταχαίως προς την ανάπτυξη του κατάλληλου επίπεδου ασφαλείας, την κατάλληλη διασύνδεση και την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh, thank you. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Να ξεκινήσουμε από τις πολιτικές ομάδες και τους εκπροσώπους τους. Ο συναδελφός Κάρινς εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Ριστόρη. Διεξοδικότατη η παρουσίασή σας και πολύ καλά μας εξηγήσατε πώς θα δραστηριοποιηθούν οι διάφοροι φορείς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Έχω μια ερώτηση και ένα σχόλιο για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα δύο ζητήματα προκύπτουν πρώτα απ' όλα οι υλικέ διασυνδέσεις και έπειτα τα ρυθμιστικά εμπόδια, η στρεβλωτική επίδραση της νομοθεσίας κάποιες φορές που δεν επιτρέπει να ενισχύσουμε τις υποδομές μας. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι πρώτον όταν ο δεύτερος κατάλογος των έργων ε, κοινή ωφελία ολοκληρωθεί. Θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας έστω περιφερειακές ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας για την αποτελεσματική διασύνδεση των κατομμύρων στο αέριο και τον ηλεκτρισμό ή θα χρειαστεί και τέτοιος γύρος. Και η δεύτερη ερώτησή μου, παρόλο που δεν είναι το θέμα μας ακριβώς σήμερα, έχει να κάνει με, το, με, τα με τους φραγμούς που υπάρχουν. Πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Θα μπορέσουμε να άρουμε τους ρυθμιστικούς φραγμούς εφόσον θα έχουμε πετύχει και τους, τις πρακτικές διασυνδέσεις. Ευχαριστούμε ο κύριος Νίκα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Ε, πρέπει να πω ότι χαίρομαι Χαίρομαι που σας γνωρίζω και σας συναντώ, αλλά λυπούμε που η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας δεν έχει αποδεχθεί τις προσκλήσεις μας να συμμετέχει σε άλλες συζητήσεις που έχουμε διοργανώσει. Λόγου χάρη συνεδριάσεις που έχουμε οργανώσει σε επίπεδο ομάδας σοσιαλιστών. Πάντως, μας δημιουργείται λίγο η εντύπωση ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας απουσιάζει. Απουσιάζει γενικώ από το διάλογο και δεν μας δίνει κάποιες σημαντικές πληροφορίες που μας είναι και απαραίτητε. Χθε ακριβώς αυτό επεσήμανα Και όταν ε, ζητάμε περισσότερα, και θα με ρωτήσεις για το πεδίο αυτό, μας λένε ότι θα έρθουν αργότερα οι απαραίτητες πληροφορίες. Θέλουμε λοιπόν μεγαλύτερο ποσοστό πράσινης οικολογικής ενέργειας και αν γίνεται και ανανεώσιμες πηγές, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Πώς μπορούμε να πετύχουμε ένα υψηλότερο ποσοστό από αυτές τις πηγές. Αρκετοί από εμά γνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα, αλλά όχι απακριβώς, θέλουμε περισσότερες πληροφορίες. Θα ήταν καλό να έρθει κάποιος και να μας πει ότι προχωρήστε για να επιδιώξετε 30% ε, ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές χωρίς να υπάρχει πρόβλημα με το σύστημα ανεφοδιασμού μας. Θέλουμε λοιπόν ακριβείς πληροφορίες σε αυτό το πεδίο σε και σε άλλα. Τι μπορούμε να κάνουμε για την καθαρή ενέργεια, δεν τα γνωρίζουμε αυτά. Η πυρηνική ενέργεια μας λένε είναι επικίνδυνη. Ο χάλιβα, ο άνθρακας, ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρξει σταδιακή εξάλληψη και θα ολοκληρωθεί που να είναι. Ε, τελικά όλοι το ίδιο ερωτώματα. Ποιο είναι το μέλλον. Τι μέλλον έχει ενέργεια σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Θέλουμε να το συζητήσουμε και με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κλάδου. Οι τιμές φύνουν. Τι θα γίνει με χώρες που δεν καταφέρνουν καν να εξασφαλίσουν τη θέρμανση για το χειμώνα. Ή τιμές ε, των ε, μπαταριών που είναι πολύ διαφορετικές από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτές λοιπόν είναι ερωτήσεις που απασχολούν όλους μας και παρουσιάσεις γίνονται, απευθυνόμαστε στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, αλλά ουδέποτε λαμβάνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε. Θα έπρεπε λοιπόν να είστε λίγο πιο δραστήριοι, λίγο πιο παρόντες. Πρέπει να μας δώσετε τις πληροφορίες που σας ζητάμε. Και έπειτα έχω και μια συγκεκριμένη ερώτηση. Η μελέτη δικτύπου για το ETS έχει ολοκληρωθεί, ναι ή όχι. E Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέ. Κύριε Γενική Διευθυντά. Ε, ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα. Ε, είναι σαφές ότι είναι περίπλοκα, αλλά και πολύ σημαντικά τα θέματα που αφορούν την ενέργεια για την Ένωσή μας. Χαίρομαι που αναφέρατε τα προγράμματα τα οποία εφαρμόστηκαν για την διασύνδεση. Ξέρω πολλά, ε, πολύ συγκεκριμένα. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποια εκτίμηση, έστω και προσεγγιστική, γιατί ξέρω πόσο περίπλοκα είναι τα θέματα αυτά. Κάποια εκτίμηση λοιπόν για το πώς είναι μεταφορές ενέργειας από το βορρά προς τον νότο. Το διατυπώνω όσο απλούστερα γίνεται. Ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας στη Βόρεια Γερμανία που θα μπορούσε να μεταφερθεί προς τα Βαλκάνια. Εάν υπάρχουν ε, οι αναγκαίες διασυνδέσεις για να βοηθήσουμε τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και θα βοηθήσουν και να αντιμετωπιστεί η αστάθεια στα δίκτυα. Πότε θεωρείτε ότι θα υπάρχει επαρκές δυναμικό ούτως ώστε χώρες όπως η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία να μην ε, αντιμετωπίσουν πρόβλημα υπερφόρτωσης των δικτύων τους, γιατί είναι οι χώρες διαμετακόμισης. Και τώρα από πλευράς των Πρασίνων, ο κύριος Έριξον. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα εγκρίθηκε η έκθεση για την οποία ήμουν εισηγητής για το στόχο του 10%. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτός ο νέος κατάλογος των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Θα ήθελα τη γνώμη σας για το κύριο θέμα που αναφερόταν στην έκθεσή μου, Εάν θέλουμε ο ποσοτικός στόχος του 10-15% να συνοδευτεί από περιφερειακούς στόχους που να εστιάζουν πολύ περισσότερο στα σημεία στένωσης σε περιφερειακό επίπεδο. Θεωρείτε ότι αυτή είναι μια σωστή προσέγγιση, θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε, θα είναι αποτελεσματική. Κάτι άλλο το λεγόμενο BAT, η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία. Πιστεύω ότι αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει τις διαδικασίες και να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις ομάδων που αντιτίθεται σε αυτά τα μεγάλα προγράμματα τα οποία εμφανίζονται και ως ασχήμια στο περιβάλλον. Μήπως μέσω λοιπόν αυτών των BAT θα μπορούσαν να επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα. Για παράδειγμα, ορισμένα καλώδια που θα μπορούσαν να είναι υπόγεια. Και τρίτον, η διαφάνεια. Βλέπω αυτό το κατάλογο των προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, PCI. Κάποια προγράμματα. Ναι, ναι, τελειώνω. Κάποια προγράμματα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα. Με εκπλήττει αυτό. Γιατί ορισμένα, όχι σαφή προγράμματα συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο. Ο κύριο Ηλικιώτη για την ΚΟΕΑ. Σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Ριστορή για την παρουσίαση του. Πράγματι τα έργα που απαρτίζουν τη δεύτερη λίζα ε, των έργων κοινού ενδιαφέροντο μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτεύξη των στόχων που έχουμε θέσει για αύξηση τη ενεργειακή απομόνωση, για ενεργειακή επάρκεια και τροφοδοσία, για αύξηση τη ενεργειακή απόδοση και μείωση τη ενεργειακή εξάρτηση τη Ένωση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα. Το ζήτημα είναι να υλοποιηθούν ε, αυτά τα έργα. Ε, κατά ρόψη μα ιδιαίτερη θετική εξέλιξη αποτελεί η υιοθέτηση έργων που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τη ηλεκτρική διασύνδεση στο Euro-Asia Interconnector ε, όπως και το East Mediterranean Pipeline. Ε, τα, αυτά τα έργα δεν συμβάλλουν μόνο στην άσκηση τη ενεργειακή απομόνωσης τη της Κύπρου και τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο στην Ευρώπη, εμεί θεωρούμε ότι είναι σημαντική και η πολιτική παρουσία μέσα από την στήριξη έργων στην περιοχή τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μια περιοχή αρκετά σημαντική και η σύνδεση πολλαπλή. Όχι, και δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο την έννοια του φυσικού αερίου, ακόμα αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση θα συνδέσει ολόκληρη την Ένωση μέσω ε, Κύπρου με το Ισραήλ και ενδεχομένω ευρύτερα στην περιοχή. Ε, θεωρούμε πολύ σημαντικές και χαιρετίζουμε αυτή τη στροφή και την, το ότι αντιλαμβάνεται σήμερα η Ένωση ότι τα νέα κοιτάσματα που υπάρχουν στην πετροχή της Ανατολική Μεροσογείου μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Για μα είναι σημαντικό να υλοποιηθούν αυτά τα έργα και αυτό που ρωτώ τον κύριο Ιστορή είναι εάν υπάρχουν ε, πέραν από τη χρηματοδότηση των μελετών ε, για αυτά τα έργα, αν υπάρχει ε, κάποιο προγραμματισμό ε, και περισσότερη σκέψη γύρω από την ε, από ένα πρόγραμμα υλοποίησης αυτών των έργων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τώρα όλοι οι άλλοι βουλευτές που θέλουν τον λόγο. Μπλάνκο Λόπεθ. Χωρίς μικρόφωνο. Ευχαριστώ για την Ιβυρική Χερσόνησο, Ισπανία, Πορτογαλία δηλαδή, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι διασυνδέσεις. Είμαι από τη Γαλλικία. Πολύ ενδιαφέρουσα η διασύνδεση της περιοχής μου. Του βορρά δηλαδή της ε, Γαλλικίας με την Πορτογαλία. Αλλά να σας ρωτήσω το εξής. Στο δεύτερο κατάλογο PCI αναφέρεται στα ισπανογαλλικά σύνορα ένα γενικό πρόγραμμα χωρίς να αναφέρεται ποια συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία θα περιλάβει η διαδρομή του. Θα ήθελα να μου πείτε γιατί δεν είναι τόσο συγκεκριμένη η διαδρομή, η χάραξη. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Ισπανία δεν θα υπερβεί το 4%. Γι' αυτό πρέπει να προωθήσουμε τέτοια στρατηγικά προγράμματα για να υπερβούμε αυτήν την ενεργητική απομόνωση της ε, χερσονήσου μας. Στην δήλωση της Μαδρίτης αναφέρονται δύο συγκεκριμένα προγράμματα μέσω των Πυρηναίων. Καντεγρή και Μαρσιλιών. Θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα τι προγράμματα προβλέπει η Κομισιόν για την περιοχή μου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Σάλφος Ζουρίνιου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, στη συνεδρίαση αυτή είχαμε πολλές ιστορικές αναφορές, είναι επέτειο για τη Ρουμανία, συγχαρητήρια λοιπόν, επίσης και η ανεξαρτησία της Πορτογαλίας το 1840 έπαυσε η κυριαρχία της Ισπανίας σε εμά, αλλά τώρα μιλάμε για την ενεργειακή Ευρώπη. Και μας ενδιαφέρει η ενεργειακή αυτοδιάθεση της Σιβηρικής Χερσονήσου. Χαιρετώ λοιπόν και εγώ τον Γενικό Διευθυντή και μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα αποτελεσματικό δίκτυο για την νέα αγορά με ανταγωνιστικές τιμές και η ενεργειακή ασφάλεια. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε πηγές ε, πόρους και επενδύσεις και η ερώτησή μου είναι η εξής. ασχοληθήκατε με το κομπικό σημείο, το hub για την Ιβηρική Χερσόνησο. Εσείς είσαστε αρμόδιος γι' αυτό. Αλλά το είδαμε και στην περίπτωση τη Γαλλία. Θέλουμε ανταγωνιστικά hub. Στην περίπτωση του Ιβηρικού hub είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά λείπουν κάποια πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, θα χρηματοδοτηθούν με το Connecting Europe Facility όσα ήδη είναι σε αυτό τον κατάλογο ή όχι. Και αν η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να συμπληρώσει κάτι από αυτά που δεν υπάρχουν στον κατάλογο όπου θα είναι σημαντική και η συνδρομή του ΕΦΣΗ. Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή όχι. Ο κατάλογος δηλαδή αυτός πώς διαρθρώνεται με δυναμικό τρόπο με τις οικονομικές ανάγκες, τις επενδύσεις που χρειάζονται στην πράξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γκύρκ. Ευχαριστώ. Καταρχάς, δύο παρατηρήσεις. Αλλά προηγουμένως να ευχαριστήσω πολύ για την εργασία που έχει επιτελεστεί στον τομέα αυτό. Δυστυχώς για πολλά προγράμματα διαπιστώνεται μεγάλη καθυστέρηση. Βέβαια για λόγους οικονομικούς, ε, Για την πρώτη ευθύνη για την ε, εφαρμογή τους τη φέρουν τα κράτη-μέλη. Αλλά θα ήθελα να καλέσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να προχωρήσουν όσο δυνατόν ταχύτερα και καλύτερα αυτά τα προγράμματα. Γι' αυτό πρέπει να, βεβαίως να κατακρίνουμε τα κράτη-μέλη. Ούτως ή άλλως ωστόσο θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, φορέων που ασχολούνται με την ε, εφαρμογή των προγραμμάτων πρέπει να βελτιωθεί. Τι σχέση έχουν για παράδειγμα τα PCI με τους περιφερειακούς καταλόγους προτεραιοτήτων. Διότι αυτοί οι περιφερειακοί κατάλογοι ε, θα έπρεπε να έχουν προτεραιότητα έναντι των γενικότερων προγραμμάτων. Αυτή είναι η πρώτη ερώτησή μου. Τι γίνεται, πώς συνδυάζονται. Και η δεύτερη ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι και αυτή έχει ένα κατάλογο υποδομών ε, προτεραιότητας. Αυτά τα λεγόμενα PCI και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει και την εκπόνηση ενός περαιτέρω καταλόγου. Τα λεγόμενα PMI, Projects of Mutual Interest, ε, αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πότε θα υποβληθεί αυτός ο νέος κατάλογος και πώς θα σχετίζεται με το κατάλογο PCI. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Κάντι. Κέλλη, συγγνώμη. Ευχαριστώ κύριε Γενική Διευθυντά. Πολύ σαφής, συγκεκριμένη παρουσίαση. Με ενδιαφέρουν λοιπόν αυτά τα PCI στα οποία αναφερθήκατε. Ιδιαίτερα αυτά που αφορούν το φυσικό αέριο. Στην εκλογική μου περιφέρεια προτείνεται ένα PCI, Sun Energy, ένα άλλο που θα μας φέρει κοντύτερα στις ΗΠΑ, που έχει στρατηγική σημασία. Ξέρω ότι ο πρόεδρος, κύριος Μπούζεκ, που πρόσφατα ήταν στις ΗΠΑ, προσπάθησε να βοηθήσει τις ενεργειακές μας εξαγωγές προς τη ΣΥΠΑ. Ερώτηση λοιπόν. Στρατηγική σημασία είναι αυτά τα προγράμματα, όχι μόνο για την Ιρλανδία, από πλευράς και εφοδιασμού και ε, διαφοροποίησης. Ε, πώς θα βοηθήσουμε να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα και από πλευράς χρηματοδότησης και από πλευράς ε, κανονιστικών ρυθμίσεων τάχιστα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Διευθυντή για τη συνεργασία μας ε, είναι το μεγαλύτερο ατού για το μέλλον και ιδιαίτερα για το GNSS ε, το Παγκόσμιο Σύστημα Πλοήγησης Μέσω Δορυφόρων. Έχουμε διάφορους φορείς, ASA, BEREC, GNS οι, οποίες, οι οποίοι φορείς ε, πρέπει οπωσδήποτε να συνεργάζονται στενά. Στην Επιτροπή ΣΤΟΑ προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε από επιστημονική πλευρά. Και έχουμε, έχουμε αναπτύξει τη στρατηγική ότι οι διάφοροι φορείς θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να μην είναι δηλαδή απομονωμένοι ο ένας από τον άλλον. Είναι πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία και για την εσωτερική αγορά ενέργειας και για την ψηφιακή αγορά και για πολλούς άλλους τομείς. Πρέπει να δούμε πώς στρατηγικά θα προετοιμάσουμε και θα ε, εφαρμόσουμε αυτή τη συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Να προσθέσω και εγώ μια ερώτηση. για το υγροποιημένο φυσικό αέριο που είναι όλο και πιο δημοφιλές όπως μας είπε ο κύριος Κέλλη και άρχισε να εξήγει και το σχιστολιθικό αέριο από τις ΗΠΑ. Έχουμε πρόσφατα προβλέψει μια ε, διεθνή αγορά αερίου. Ε, κάτι που δεν προβλεπόταν ως τώρα, μόνο για το πετρέλαιο υπήρχε το ανάλογο, όχι για το φυσικό αέριο. Τι θα γίνει με τους σταθμούς παραγωγής ενέργειες και τον κατάλογο και τι θα γίνει και με τη γεωγραφική κατανομή. Συγγνώμη, ξέχασα τη λέξη, αλλά καταλάβατε τι εννοώ. Μπορείτε να ξεκινήσετε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι το υγροποιημένο φυσικό αέριο, Ξέρετε πώς έχει κατάσταση. Υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις από ηλική σκοπιές στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε μερικά σημεία στην Γαλλία. Αλλά χτίζουμε και νέε εγκαταστάσει, δημιουργούμε νέε διασυνδέσει εκεί που υπάρχουν αυτές οι πραγματικέ εγκαταστάσει, για να υπάρξει ευκολότερη πρόσβαση στο αέριο και διαφοροποίηση. Αυτό είναι απολύτως το σημασία τη στιγμή που έχουν γνωρίσει μια επανάσταση στην ε, αγορά του αερίου, με φοβερέ ταχύτητε, με νέου παραγωγού, Όχι μόνο τι ΗΠΑ, όχι μόνο την Αυστραλία, τον Καναδά, αλλά και αφρικανικές χώρες με ανακαλύψεις, την Αίγυπτο λόγου χάρη. Πέραν αυτών που ήταν ήδη γνωστά ως κοιτάσματα στην Αλγερία. Γνωρίζουμε λοιπόν και αποφελούμαστε από όλα αυτά, εννοώ τις νέες υποδομές ε, για τις διασυνδέσεις και τους ε, σταθμούς παραγωγής και προσπαθούμε να στηρίξουμε την διαφοροποίηση και την ανταγωνιστική αγορά. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να υποστηριχθούν κάποια έργα. Ακόμη και για τις πιο ευάλωτες περιοχές όπως η Κροατία, η Πολωνία ή οι χώρες της Βαλτικής. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σημείο, τις πραγματικές διασυνδέσεις και τα ρυθμιστικά εμπόδια. Για τις διασυνδέσεις είπα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του δεύτερου καταλόγου. Για να φτάσουμε για το αέριο το 10% διασύνδεσης παντού. Η Κύπρος και η Ισπανία θα ακολουθήσουν όπως είπα. Αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα για το αέριο. Για το αέριο. Όχι για την ηλεκτρική ενέργεια. Όχι. Για την ηλεκτρική ενέργεια είναι το 10% για να ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Θα πρέπει να πετύχουμε αυτό το στόχο προτεραιότητα. Και αυτό δεν είναι μόνο πολιτικό, από πολιτική σκοπιά σημαντικό, αλλά είναι σημαντικό για να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει και η σωστή ροή ενέργεια από βορρά προ νότο και από ανατολή προ δύση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα αναπομέναντα σημεία συμφόρησης. Τώρα ως προς τους ρυθμιστικούς φαγμούς. Πράγματι δεν μπορούμε να δράσουμε ε, στις πραγματικές πτυχές χωρίς να αντιμετωπίσουμε τα ρυθμιστικά θέματα. Γι' αυτό λοιπόν η επιβολή της υπάρχουσας νομοθεσίας είναι πρώτη σημασία. Αλλά και το να υπάρξει κάποια εξέλιξη, κάποια πρόοδος Γι' αυτό ως το τέλος της ερχόμενης χρονιάς θα παρουσιάσουμε μια σημαντική νέα πρόταση που θα αφορά τη νέα ε, δομή της αγοράς. Ένα νέο σύνολο κανόνων προκειμένου να επιταχυνθεί η νομοθετική ε, προσπάθεια και να ε, εδρεωθεί η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα. Αυτό αφορά λόγω χάρη θέματα όπω η αποθήκευση. Δεν είναι σίγουρα η κατάσταση που είχαμε πριν από 30 χρόνια. Πριν από 30 χρόνια δεν είχαμε 27% ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Το θέμα τώρα είναι πώς θα διαχειριστούμε τις διακυμάνσεις αυτή τη στιγμή για να έχουμε και απόθεμα. Ε, σε αυτήν τη λογική λοιπόν η αποθήκευση θα είναι μια από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Συμφωνώ στο παρελθόν η αποθήκευση είχε υποτιμηθεί. Είχε υποτιμηθεί στην προσέγγιση μας. Αυτό θα αλλάξει και για αυτό ακριβώς μέσα από την πρότασή μας με καλύτερο σχεδιασμό θα αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση για να βεβαιωθούμε ότι αυτό που είναι ζωτικής σημασίας θα μας επιτρέψει να σταθεροποιήσουμε το δίκτυο. και θα υπάρξει, θα αντιμετωπίσουμε την τόσο γοργά εναλλασσόμενη παραγωγή ενέργειας, διότι το 2020, ξέρετε ότι πάνω από 50% της ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό απαιτεί νέους κανόνες, αλλά και νέα μέσα, προκειμένου να ανταποκριθούμε. Δεν, θα, ε, δεν έχουμε μπροστά μας μια αγορά ε, απαράλλαχτη και ακίνητη. Πρέπει να τακτοποιήσουμε ταυτόχρονα και τις νομοθετικές πτυχές και το τι γίνεται στην πράξη και τις τεχνολογικές λύσεις. Γι' αυτό όλα αυτά λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία. Πώς να ε, βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξουν οι κατάλληλες διασυνδέσεις για το ευρωποιημένο φυσικό αέριο και από βορρά προς νότο και θα αντιμετωπίσουμε και τις χρελίδες στην αγορά και πώς θα αντιμετωπίσουμε το blackout ή κάποιο έλλειμμα στην ε, ε, προμήθεια. Αυτό θα είναι επίσης μια μεγάλη πρόκληση και γι' αυτό θα απαιτηθεί η διαρκής και μόνιμη συνεργασία μεταξύ των ε, φορέων ε, διαχείρισης του δικτύου, του δικτύου διανομής και των ρυθμιστών. Διότι πρέπει να ξεπεράσουμε το σημερινό επίπεδο διακρατικού εμπορίου για το αέριο και τον ηλεκτρισμό. Θα χρειαστεί νέα διασυνοριακή διαχείριση. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλες τις νέες τεχνολογίες. Αλλά να ε, οδηγήσουμε και στα σταθεροποίηση του δικτύου ακόμη και όταν έχουμε ε, εχμή στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του επίπεδου ενέργειας και των δοκιμάσεων που είναι υπολόγιστες απολύτως ε, σοβαρό αυτό. Επίσης, όπως είπα, η αντιμετώπιση των σημείων συμφόρηση, η αξιοποίηση των τεχνολογικών λήψεων και λύσεων και όσο αφορά την διαφάνεια. Το ανέπτυξα νομίζω και πραγματικά ικανοποιούμε ιδιαίτερα για κάποιε νέε πρωτοβουλίε που στηρίζουμε. Λόγω χάρη η νέα προσέγγιση που ομαδοποιεί κάποιο στοιχείους σημαντικούς TSO και NGO. Τους διαχειριστές δικτύου μεταφοράς Εδώ ε, έχουμε κάνει τέτοιες ενέργειες στην Ισπανία και αλλού. Και ο στόχος είναι να εξηγήσουμε γιατί κάποια από αυτά τα έργα θα είναι υποφελή όχι μόνο προς την ασφάλεια Το είπαμε στο νέο φόρουμ, στο πρώτο, στις πρώτες συζητήσεις του φόρουμ ε, για τις νέες υποδομές ενέργειας στην Ευρώπη. Ήταν και ο κύριος Έριξον και ο κύριος Πέτερσον. Αλλά θα είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της ε, συνεργασίας των TSO στο μέλλον θα αποτελέσει ενδεχομένω το αντικείμενο νέου κανονισμού, διότι θα υπάρξει κερδοφορία, αυξημένη αξία. και ως προς την ασφάλεια και ως προς την συμμετοχή στο δίκτυο των ε, πηγών των ανανεώσιμων. Εδώ μετά θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι οι καλύτερες εναλλακτικές για να προχωρήσουμε. Όμως, ό,τι επιλογή και να κάνουμε θα πρέπει να είναι διαφανής και ε, κυρίως να εξηγηθεί κατά το στο ευρύ κοινό για να αντιμετωπίσουμε τις εναπομείνασες αντιστάσεις. Σε ό,τι αφορά τα επικουρικά προγράμματα, Μερικέ φορέ η σημασία κάποιων προγραμμάτων για κάποιε περιφερειέ, γεωγραφικέ περιοχέ είναι δύσκολο να γνωριστεί ε, αν δεν υπάρχει ε, επαρκής οριμότητα. Είναι δύσκολο να το πιστεί το πλέον σημαντικό έργο που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την ε, πολυπόθητη διαφοροποίηση. Έχουμε και τα διδάγματα έχουμε αντλήσει το παρελθόν που είναι σημαντικά για να αποτιμήσουμε σωστά το τι θα κάνουμε στο μέλλον βάσει των πορισμάτων των μελετών που έχουμε ως τώρα στα χέρια μας. Και με τα μεγάλα ποσά ε, χρηματοδότηση που διαθέτουμε, κυρίως από την ε, διευκόλυνση για τη διασύνδεση της Ευρώπης. Επί της αρχής, η επιστροφή των επενδυτών στα η απόδοση των επενδύσεων στα ενεργειακά έργα είναι κάτι που επιστρέφει, αλλά είναι και κάτι που καλύπτουν συνήθως οι χρήστες. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες, όπως την διευκόλυνση για τη της Ευρώπης, με κάποια μέτρια ποσά, ε, κάθε δισεκατομμυρίων ευρώ για ολόκληρη την περίοδο, αλλά θα αξιοποιήσουμε και άλλε δυνατότητε όπω τα διαφορετικά ταμεία, όπω η στήριξη τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή του, ε, Ευρωπα... του τα... Ευρωπαϊκού Ταμείου για τι Στατικέ επενδύσει. Εκεί ξέρετε ότι υπάρχουν τρει προτεραιότητε: υποδομέ ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια και αέριο, τι διασυνδέσει του πρώτα, μεγάλα έργα για του ανανεώσιμε έπειτα και ε, σχέδια ενεργειακής αποδοτικότητα. Αυτέ είναι οι τρει προτεραιότητε που έχουμε θέσει. σε ό,τι αφορά την διασύνδεση Πορτογαλία. είναι άκρο σημαντικό και θα ξέρετε πολύ καλά πόσο πρόεδρος έχει γίνει ως τώρα. Πρέπει να πω ότι η Καμπή ήταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου 2013 με το νέο ενεργειακό πλαίσιο ως το 2030. Τότε πραγματικά φτάσαμε σε μια πολιτική συμφωνία στο υψηλότερο επίπεδο όπου η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Γαλλία συνεννοήθηκαν Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για να ολοκληρωθεί το ΙΝΕΒ, αλλά και να καθορίσουμε τη θετική μας ε, των ε, διαχειριστών του δικτύου δυναμής με τη συμμετοχή τουλάχιστον των τριών αυτών χωρών στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο όπως είπα και κατά συνέπεια θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την υλοποίηση του προγράμματος δράσης συμπεριλαμβανομένων των δύο έργων που διαπερνούν τα Πυρηναία. Και επίσης και του έργου που περνάει από τον ε, Βυσκαϊκό. Την ε, περασμένη Δευτέρα μιλήσαμε με την ε, Εκδοστική Επιτροπή της Ραντελέκτρικα για να βεβαιωθούμε ότι η υλοποίηση θα γίνει γοργά και θα δοθεί απαραίτητη προσοχή για να υπάρξει απαραίτητη πρόοδος σε όλα τα μέτωπα. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά έργα, αλλά και όταν μιλάμε για νέα έργα, νέες δυσυνδέσεις, όπως Ισπανίας Μαρόκου ή Πορτοκαλίας Μαρόκου. Άκρος σημαντικό, με τη δική μας πολιτική στήριξη. Επίσης, θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ε, υλοποίηση και την μείωση των περιορισμών των καθυστερήσεων. Το είπατε κι εσείς, κάποιες φορές τα κάτι μέλη φταίνουν για τις καθυστερήσεις, όμως καθησυχάζομαι επειδή έχουμε πλήρη στήριξη από όλα τα κάτι μέλη ως προς την προετοιμασία ενός, την εκπόνηση ενός καταλόγου σε επίπεδο γεωγραφικών περιοχών που θα πρέπει να είναι έτοιμο ότι θα έχουμε την τελευταία συνάντηση με τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και χάρηκα πολύ με αυτό που είπε και ο κύριο Ρούμπιχ. Αυτό το είδου συνεργασία στην Ευρώπη είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία και επειδή και ωφέλη θα φέρει, το είπε και ο κύριο Κέλλη, ωφέλη οικονομικά αλλά και θα στηρίξει την αλληλεγγύη. Το είδατε και το γνωρίζετε πολύ καλά. Η διασύνδεση και υποδομές της ξεπερνά τον τομέα της ενέργειας. Φέρνει τα κάτι μέλη και τους πολίτες τους πιο κοντά. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Γενική Διευθυντά. Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σας και πολύ λεπτομερής. Χρειαζόμασταν κάτι τέτοιο, διότι έργα σημαίνει πράξη. Ίσως αν είχαμε άλλο χρόνο να μας δίνετε και άλλες λεπτομέρειες, να κρατούσε άλλη μία ώρα η συνεδρίασή μας, δεν έχουμε όμως δυστυχώς άλλο χρόνο. Ήθελα να ευχαριστήσω και τους ε, διερμηνείς μας που βρισ... έμειναν μαζί μας περισσότερα από ό,τι προβλεπόταν. Συνάδελφοι, θυμίζω σε όλους μας και παρακαλώ θυμηθείτε το στις 3, έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΙΜΚΟ για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Και θα βρεθούμε όλοι εδώ σε αυτή την αίθουσα στις 3 το απόγευμα. Δεν είναι και πολύ μεγάλο το διάλειμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά.